Mes chers collègues, pour ceux Λοιπόν, όσοι είναι εδώ τους ευχαριστώ για την παρουσία τους. Θα επανέλθουμε λοιπόν στη συνεδρίασή μας και θα ενδιαφερθούμε με τις διαφορές στην ε, πρόσβαση των ε, φαρμακευτικών προϊόντων στις ευρωπαϊκές αγορές. Euh, euh, Θα σας δώσω το λόγο λοιπόν στον κύριο Καναβό. Θα μας παρουσιάσει το θέμα. Και υπάρχει χρόνος, μπορείτε να παρουσιάσετε με άνεση το θέμα σας. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε. Να σας παρουσιάσω το έγγραφο το οποίο ασχολείται με τις διαφορές το κόστος πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση των προϊόντων αυτών. Ελπίζω να έχετε όλοι το φάκελο μπροστά σας. Θα σας περιγράψω κάποιες από τις διαφάνειες Εξετάζοντας τις ε, τα στοιχεία τα οποία μας είχατε δώσει όταν μας ζητήσατε να κάνουμε την παρουσία, προσπαθήσαμε να εξετάσουμε τους λόγους για τους οποίους ποικίλουν οι τιμές των προϊόντων ε, στα διάφορα σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασχοληθήκαμε με τα ποσοστά δαπανών για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, και να ασχοληθούμε επίσης και με το θέμα της παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και έρευνας και να μας επιτρέψετε να κάνουμε για κάποιες συστάσεις σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα δείτε στο φάκελο που έχετε μπροστά σας κάποιες από τις διαφορές που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε σχέση με το ΑΕΠ, οι οποίες δεν αντικατοπτρίζονται ένα προς ένα, στον τομέα των δαπανών για την υγεία κατά κεφαλήν, όπως επίσης και των δαπανών για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Αν τα εξετάσει κανείς με δυναμικό τρόπο υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις διάφορες χώρες της Ένωσης. Το θέμα είναι σε τι οφείλονται οι διαφορές αυτές. Αυτό μας οδηγεί στο θέμα και των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων. Παρατηρώντας την κατάσταση διαπιστώνει κανείς διαφορές στα φαρμακευτικά προϊόντα και για λόγους προέλευσης αλλά και για διαφορετικούς λόγους. Οι διαφορές αυτές μπορεί να έχουν πολύ μεγάλο ύψος. Ακολουθούνται διαφορετικές διοντολογίες, διαφορετικές μελέτες, ε, οι οποίες έχουν γίνει στο παρελθόν γύρω από το θέμα και επί τη βάση συγκεκριμένων αποδείξεων καταλήγουμε σε κάποιες προσπάθειες που έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο και που ζητούν για ένα καλάφι συνταγών που δικαιολογεί και εξηγεί τις διαφορές των τιμών από τη χαμηλότερη στην υψηλότερη κατά 25 περίπου τις 100 όπως επίσης και διαφορές στις τιμές ανάμεσα στο ευθυνότερο και το ακριβότερο κράτος μέλος, που φτάνουν στο 41%. Σε ορισμένες περιπτώσεις και για όχι πρωτότυπα αλλά γενικ... Ε, ε, προϊόντα higher. Um, in some cases they can be significant. προϊόντα. Ε, οι διαφορές αυτές είναι πολύ χαμηλότερες ανάμεσα στις διάφορες χώρες. Ο φαρμακευτικός τομέας είναι σημαντικός εργοδότης στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντιπροσωπεύει περίπου το 3,5% της συνολικής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της παρασκευής και συνεισφέρει και στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης και δεν συμπεριλαμβάνει μόνο τα πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα αλλά και τα δευτερευόντως τα γενώσιμα τα οποία συνεισφέρουν στην ευρέωση της βιομηχανικής βάσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλες οι διαφορές ποικίλουν πολύ μεταξύ τους και γι' αυτό απαιτούνται κάποιες εξηγήσεις. Αν προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες τέτοιες εξηγήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να δούμε κάποιες πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται σε επίπεδο εθνικών κρατών. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα διακανονιστικά πλαίσια, να εξετάσουμε την τιμολόγηση και τις επιστροφές του κόστους των φαρμακευτικών προϊόντων. Τα πλαίσια αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη η τιμολόγηση των φαρμάκων ρυθμίζεται κεντρικά στις περισσότερες χώρες, υπάρχουν όμως διαφορές σε σχέση με την αναφορά των τιμών, υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι στην αξιολόγηση του ύψους της τιμής, κάτι το οποίο εξηγεί τις διακυμάνσεις των τιμών. Αυτό οφείλεται και στην προσφορά επίσης, αν δει κανείς ε, ιδιαίτερα ε, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα. Υπάρχουν βέβαια ε, Υπάρχουν στοιχεία που μας επασχολούν στον τομέα όχι μόνο της προσφοράς αλλά και στον τομέα της ζήτησης. Δοτίθεται σε συζήτηση η συμπεριφορά των συνταγογραφών των ιατρών όπως επίσης και η συμπεριφορά η καταναλωτική των ασθενών. Ε, σχετικά με τη συμπεριφορά των γιατρών οι οποίοι συνταγογραφούν Υπάρχει μια τάση να πιεστούν να συνταγογραφούν γενώσιμα προϊόντα και επίσης να πιστούν και οι φαρμακοποιοί να χορηγούν τέτοιου είδους προϊόντα. Όλες αυτές λοιπόν οι πολιτικές και όλα αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο και με διαφορετική ένταση στα διάφορα κρατημέλη. Το πάζολ λοιπόν γίνεται ακόμα πιο περίπλοκο, ακόμα πιο σύνθετο, γιατί πέραν όλων όσων είπα, οι διαφορετικές διακανονιστικές ρυθμίσεις αφορούν και την αλυσίδα διανομής των προϊόντων και σε επίπεδο χονδρικής και σε επίπεδο λιανικής. Κάτι το οποίο δεν είναι κάτι που προκαλεί επιπλέον κόστος, αλλά παρόλα αυτά συνεισφέρει πολύ στις συνολικές δαπάνες για τα φαρμακευτικά προϊόντα. Βλέποντας λοιπόν τι γίνεται και σε επίπεδο προσφοράς και ζήτησης, διαπιστώνει κανείς ότι η συνεισφορά στο κόστος της αλυσίδας διανομής είναι σχετικά υψηλή. Και τίθεται εδώ και το θέμα των φορολογικών δομών του ΦΠΑ, το ύψος του ΦΠΑ που σε ορισμένες χώρες είναι 0 και φτάνει το 25% για συνταγογραφούμενα προϊόντα σε άλλες περιπτώσεις. Κάποιες από αυτές τις ε, κρατικές ή διακανονιστικές ρυθμίσεις έχουν οδηγήσει σε ορισμένα προβλήματα πρόσβασης σε ορισμένα τμήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, το αν αυτά τα προβλήματα πρόσβασης των προϊόντων οφείλονται στις διαφορές ε, μεταχείρισης των συγκεκριμένων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της τιμολόγησης των προϊόντων ανακράτος μέλος, και της αξίας την οποία παρέχει η χρήση των συγκεκριμένων μεθοδολογιών είναι κάτι το οποίο μένει να καθοριστεί. Μπορεί όμως η διαφορά στη μεθοδολογία να οδηγήσει σε διαφορές ε, για τη διάδοση ορισμένων τεχνολογιών τέτοιου τύπου στις διάφορες χώρες. Σε ορισμένες μικρές χώρες, σε μικρά κρατημέλη, Έχουμε και το θέμα της μικρής αγοράς βέβαια, του μεγέθους της αγοράς και γι' αυτό ορισμένα προϊόντα ίσως και να μην είναι καν διαθέσιμα ή όταν είναι διαθέσιμα να είναι πάρα πολύ ακριβά και κάποια από τα γενώσιμα να μην είναι καν διαθέσιμα επίσης. Επίσης υπάρχει και το θέμα της διασύνοριακής εμπορίας φαρμάκων, φαρμακευτικών ουσιών, η οποία κάνει το λεγόμενο διαιτητή, το οποίο οφείλεται στο λεγόμενο διαιτητικό φαινόμενο, δηλαδή εξάγονται προϊόντα από μια χώρα που έχει χαμηλές τιμές προς μια χώρα η οποία έχει υψηλές τιμές. Αυτό παραδοσιακά οδηγεί σε διαφορές τιμών από 1 μέχρι 20% και καλύπτει και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανάλογα με την περιοχή που κυμαίνεται και αυτό. Υπάρχουν πολλά θέματα λοιπόν τα οποία αφορούν την πρόσβαση των προϊόντων οφείλονται στα διαφοροποιούμενα διακανονιστικά ε, καθεστώτα που ισχύουν ανάλογα σε κάθε χώρα. Τα εξετάζουμε στην έκθεσή μας όλα αυτά. Σχετικά τώρα με τη δυνατότητα επιλογών. Οι επιλογές αυτές οφείλονται και, στα, και οφείλονται, μάλλον μπορούν να ασκηθούν και από το εθνικό επίπεδο και από το κοινοτικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο λαμβάνονται υπόψη οι διακανονιστικές πρακτικές σε επίπεδο κρατών μελών. Έχει σημασία να συνεχίσουμε να αξιολογούμε συστηματικά την πολιτική στον τομέα των φαρμάκων, να βλέπουμε επίσης τις επιδόσεις των κρατών μελών σε οικονομικό επίπεδο, αλλά δεν εξετάζουμε πάρα πολύ συχνά τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων μέτρων τα οποία εφαρμόζονται. Είναι σημαντικό να γίνει κάτι τέτοιο και αν δεν το κάνουμε επαρκώς πρέπει να γίνει πλέον. Υπάρχουν λοιπόν θέματα όπως και οι ε, μεθοδολογίες ε, διαμήρασης κινδύνου σε σχέση με το τι είναι ωφέλιμο, τι δεν είναι ωφέλιμο, πώς μπορούμε να μεγιστοποιήσουμε τις ωφέλιμες μεθοδολογίες. Υπάρχει επίσης και μια έκκληση γενικότερη για την αύξηση της χρήσης γενώσιμων προϊόντων, γιατί θεωρούνται ωφέλιμα και σε επίπεδο δημοσιονομικό και στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Σε ορισμένες χώρες το ποσοστό των γενώσιμων είναι ιδιαίτερα υψηλό, σε άλλες χώρες πάλι είναι ιδιαίτερος χαμηλό. Και αυτό οφείλεται στο μείγμα της πολιτικής το οποίο ακολουθείται κατά περίπτωση. Έχει σημασία λοιπόν να συνεχίσουμε να δίδουμε κίνητρα προς την καινοτομία στον τομέα αυτό των φαρμακευτικών προϊόντων γιατί όχι μόνο αυτό είναι κάτι το οποίο επιτρέπει να μείνουν σε ζωή οι έμποροι που ασχολούνται οι παροχής, αλλά και βοηθά και τους ασθενείς να την χάνουν καλύτερης θεραπείας και όχι μόνο ποσοτικά, αλλά και να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής τους. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα έχει σημασία να συνεχίσουμε τις προσπάθειες που έχουν αρχίσει να υπάρξει περαιτέρω ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ανταλλάσσουμε τις εμπειρίες μας, να ξεκαθαρίσουμε το τι πηγαίνει καλά και τι όχι στις διάφορες χώρες μέλη. Να συνεχίσουμε τις προσπάθειες επίσης τη ενθάρρυνση τη καινοτομία στον τομέα των βιοδυναμικών στι διάφορε χώρε να συνεχίσουμε την ενθάρρυνση της καινοτομίας γενικότερα και από την άλλη πλευρά του φάσματος να ενθαρρύνουμε τη χρήση των γενώσιμων προϊόντων και στο σύνολο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν προβλήματα που αφορούν κάποιες πολύ μικρές αγορές, τα οποία επίσης θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και τέλος, σε επίπεδο ε, εμπορίας ε, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η πρακτική και σε επίπεδο αρχής και επί της ουσίας και να ενθαρρύνουμε περαιτέρω έρευνες και συζητήσεις για τις πρακτικές οι οποίες ακολουθούνται. Αυτό αφορά την αλληλοεπίδραση ανάμεσα στην ενιαία αγορά και τις επιμέρου εθνικές πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο βέβαια να παρουσιάσει κανείς με επαρκή τρόπο σε 10 λεπτά ένα θέμα το οποίο αφορά τόσο πολύ κόσμο. Σας έδωσα όμως ένα μικρό δείγμα του τι περιλαμβάνεται στο έγγραφο και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτή την σύνθεση την οποία κάνατε της εκθεσή σας, πάρα πολύ πλούσια και σε ένα θέμα το οποίο μας αφορά όλους και από πολύ κοντά. Θα δώσω λοιπόν τώρα το λόγο στους πρώτους συναδέλφους που το ζήτησαν, στον κύριο Σνέλχαρτ πρώτα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα τη μελέτη αυτή που δώσαμε εντολή να συνταχθεί και έχω υπόψη διαβάζοντας την μπορεί κανείς να κερδίσει με επισκόπηση ποια προβλήματα υπάρχουν και ποιες λύσεις προτείνονται. Ωστόσο όμως έχω προς τον συντάκτη κάποιες ερωτήσεις που θέλω να θέσω και που για την άποψή μου για την ολοκλήρωση της μελέτης, δηλαδή κύριες πηγές, για τέτοιου είδους μελέτες και γνωρίζουμε ότι στη μελέτη σας είχατε ε, τοποθετηθεί για συγκεκριμένα θέματα και χρησιμοποιήσατε και στοιχεία του Συλλόγου των Φαρμακοποιών. Όχι όμως ε, σε σχέση με τους ε, μεγαλεμπόρους, τους, τις μεγάλες αποθήκες, τους άλλους εμπόρους ή σε εισαγωγικά αντικειμενικές πηγές μεταξύ άλλων. Ερώτηση τέτοιου είδους ε, μελέτες που καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα όσον αφορά τον ε, συντάκτη της έκθεσης και παράλληλα με εκθέσεις που αφορούν εισαγωγές φαρμάκων λαμβάνονται υπόψη ή όχι. Δεύτερη ερώτηση σε σχέση με τα προβλήματα των οθευμένων φαρμάκων. Αναφέρεται εδώ ότι αυτές, οι παράλληλες εισαγωγές φαρμάκων αποτελούν κίνδυνο. Τώρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο τον Φεβρουάριο του 2011 η φέτος έθεσε σαφείς αποφάσεις που έλαβε και ακριβώς αυτή η εισαγωγή νοθευμένων φαρμάκων είναι κάτι που θέλουμε να αποφύγουμε και να παρεμποδίσουμε που ισχύουν και για το παράλληλο αυτό εμπόριο. Και αυτά δεν τα βρίσκω στην έκθεσή σας, αυτές τις αποφάσεις μας, αυτά τα στοιχεία. Η τρίτη παρατήρηση, κατά την ανάγνωση της μελέτης, της ε, μελέτης αυτής, καταλήγω αμέσως στο συμπέρασμα ότι η σχέση σε σχέση με τους ε, ε, ασθενείς και για την αγορά φαρμάκων. Οι μεγαλέμποροι όμως και οι φαρμακοποιοί έχουν την, τον ρόλο να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών με φάρμακα. Χωρίς αυτούς δεν μπορούν οι ασθενείς να αποκτήσουν φάρμακα ποιο είναι το είδος ε, ε, του ανεφοδιασμού που φαντάζεται ο συντάκτης ότι θα έπρεπε να ακολουθηθεί ώστε όλοι οι ασθενείς να έχουν ποιοτικά αναβαθμισμένα και ασφαλή φάρμακα στη διάθεσή τους. Αυτές οι τρεις ερωτήσεις. Θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να τοποθετηθείτε. Και πιστεύω ότι υπάρχει εδώ ένα κενό που πρέπει να καλυφθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. όπως είπε και ο κ. Σνέλχαρτ, ε, χωρίς να έχω διαβάσει επιστολές από ε, φαρμακευτικές εταιρείες. Για μένα δεν μου προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι τα κύρια αποτελέσματα σελίδα 32, ιδιαίτερα για, τους, ε, για τα ζητήματα παράλληλου εμπορίου. Εκεί βλέπετε τη σύγκριση των τιμών, που ούτε αυτό μου με ξένησε, ότι δηλαδή τα φαρμακευτικά είδη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που βέβαια συμμετέχουν σε αυτό το παράλληλο εμπόριο, αλλά και τα γενώσιμα φάρμακα, άμα το δείτε αυτό, έχουν τετραπλάσια τιμή σε σχέση με τα γενώσιμα φάρμακα. Αυτό μας δίνει μια ιδέα για το τι συμβαίνει. Για τα ζητήματα πολιτικής, δεν ε, είμαι σίγουρη ότι κατάλαβα καλά. Ε, γιατί και εμείς τώρα εξετάζουμε εδώ και καιρό την νομοθεσία ε, στον τομέα ε, των φαρμάκων. Ε, ίσως θα ήταν περισσότερο ακαδημαϊκού επίπεδου συζήτηση στο, στο LSC. Αναφέρατε το ε, επίπεδο απασχόλησης στον ε, τομέα της φαρμακομιομηχανίας. Συμφωνείτε μαζί μου ότι ο παράγοντας της απασχόλησης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στην αρχική παραγωγή, δηλαδή και στον τομέα της έρευνας ε, ε, περισσότερο στα προϊόντα ε, με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρά στα γενώσιμα. Αν συμφωνείτε μαζί μου και πιστεύω ότι θα συμφωνείτε, δεν ξέρω αν εγώ συμφωνώ μαζί σα για την δυνατότητα επιλογή πολιτική σε εθνικό επίπεδο για την αύξηση των γενώσιμων φαρμάκων. Γιατί αυτό για μένα θα αποτελούσε αντίφαση γιατί αφενός υπογραμμίζεται ε, τον παράγοντα της απασχόλησης στην φαρμακομηχανία και αφετέρου θέλετε να αυξήσετε το μερίδιο των γενοσύμων. Ε, κάτι που θεώρησα ενδιαφέρον ήταν ε, το τμήμα που αναφέρεται στο HTA. Ε, σίγουρα θα έχετε παρακολουθήσει τον διάλογο για την διασυνοριακή περίθαλψη και είδατε τι ε, ε που αντιμετωπίσαμε. Αν βλέπετε πώ μπορούμε να, να πείσουμε τα κράτη-μέλη, όπω το Μενό Βασίλειο αλλά και άλλου, να έχουν... Να, ε, να ανταλλάσσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ε, βέλτιστες πρακτικές τους στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό θα μας βοηθούσε ιδιαίτερα, γιατί δεν έχουμε πλέον νέες ιδέες. Μετά, τις ε, επιλογές πολιτικής ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και, και πάλι θέλετε την περαιτέρω διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων των πρακτικών, ε, αυξημένου συντονισμού. Θα ήθελα να ακούσω τις ιδέες σας. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί δυστυχώς... η φαντασία μου δεν με επιτρέπει άλλες ιδέες προς το παρόν. Δεν είμαι σίγουρη όταν αν δεν υπάρχει, συμφωνείτε μαζί μου ότι αν δεν υπήρχε ε, συνταγογραφούμενο φάρμακο με, με δίπλωμα ευρεσιτεχνία αρχικά, μετά δεν θα μπορούσε να υπάρχει γενώσιμο φάρμακο. Επομένω, πώ πιστεύετε ότι πρέπει να αυξηθεί η έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη, ίσω να είναι ε, να μην το κατάλαβω καλά. Αλλά για μένα η, απλώς η αύξηση των γενοσύμων ε, δεν έχει νόημα όταν δεν υπάρχει προηγουμένως φάρμακο το οποίο προστατευόταν από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Για κάποιες από τις επιλογές, ε, τις πολιτικές επιλογές εδώ συμφωνώ. Εντάξει, δεν έχει τίποτα κακό η πρότασή σας, αλλά ίσως είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Πώς δηλαδή θα δώσουμε ε, κίνητρα στα, ε, στα κράτη-μέλη να συντονίσουν ε, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης τους όταν δεν είναι διατεθειμένα να το κάνουν προς το, προς το παρόν. Ευχαριστούμε, Καρς Yeah, ε, for... Ευχαριστούμε για αυτή την έκθεση. Αυτό που με εκπλήσει είναι η ε, σημαντική αύξηση του κόστου των φαρμάκων από το 2000 στο το 2008 σε αρκετές χώρες. Γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ακολούθησε το ίδιο πρότυπο, ε, έκαναν κάτι ιδιαίτερο εκεί κάτι ξεχωριστό. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Μήπως μπορούμε να αντιλήσουμε κάποιο παράδειγμα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Κάτι άλλο για το πολύ χαμηλό επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης ε, 15 με 20%. Πολύ χαμηλό μερίδιο λοιπόν του κόστους πάει στην έρευνα. Στις προτάσεις σας, μου λείπει μία πρόταση, κάτι που θα συζητηθεί αύριο στη Γερουσία των ΗΠΑ, τα, κονδύλια κόστους είναι ένας εναλλακτικός μηχανισμός χρηματοδότησης ε, ε, τη έρευνα. Ε, προσδιορίζουμε τις προτεραιότητε στην υγεία, λέμε ποια είναι τα φάρμακα που χρειαζόμαστε περισσότερο και μετά τα κοστολογούμε. Ίσως σε μικρά τμήματα. Για παράδειγμα έχουμε ένα για τη διαγνωστική και ούτω καθεξής. Αλλά ε, τα κοστολογούμε και μετά όλη η παραγωγή απελευθερώνεται από τις άδειε. Και έτσι δεν χρειαζόμαστε αυτή την παράλληλη εισαγωγή, ε, ούτε το πρόβλημα των... Ε, παραποιημένων φαρμάκων, γιατί το όριο κέρδους είναι πολύ μικρό. Την έχετε εξετάσει αυτή την ελλακτική λύση και επιλέξατε να μην τη συμπεριλάβετε στην έκθεσή σα ή μήπω δεν το έχετε εξετάσει καθόλου. Ευχαριστούμε. Πίτερ Λίζα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να προσθέσω τη φωνή μου στην ερώτηση του κυρίου Χορσνέρχαρτ για τις παράλληλες εισαγωγές φαρμάκων. Αυτή ήταν ουσιαστικά η αφορμή γιατί αποφασίσαμε να ζητήσουμε να συνταχθεί μια μελέτη για λογαριασμό μας. Διότι στη συζήτηση για την όθευση φαρμάκων θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι και αυτό θα ήταν μια αφορμή για νόθευση φαρμάκων. Και αυτό θα ήθελα και εγώ να ε, τύχει συνέχεια. Και είπαμε, εφόσον υπάρχουν τόσο τεράστιες διαφορές τιμών, όταν και εφόσον υπάρχουν, το παράλληλο εμπόριο μπορεί να καταστήσει μικρότερες αυτές τις διαφορές, να τις απαμβλύνει. Ερώτηση, ποιος κερδίζει άμεσα από το παράλληλο εμπόριο ή έμποροι. Έχουμε όμως και έμεσες επιπτώσεις όταν υπάρχει παράλληλο εμπόρευμα. Δεν είναι μόνο η απάμβληση των διαφορών τιμών σε σχέση με κάποιους ε, επιχειρηματίες ε, και δεν είναι απόλυτη η εξίσωση. Δεν είναι τόσο σαφές και δεν είναι εύκολο να υπολογιστούν όλα αυτά επακριβώς όταν μόνο στρέφει το βλέμμα κανείς προς μία κατεύθυνση και δεν βλέπει προς την άλλη όταν υπάρχει για παράδειγμα ο ανταγωνισμός και διαμορφώνει τις τιμές αντίστοιχα. Δεύτερο σημείο και θα ήθελα να σας παρακαλέσω αν μπορείτε να πείτε κάτι γι' αυτό για τα κόστη των διαφορετικών συστημάτων. Έχουμε εκατοντάδες στελέχη στις μεγάλες επιχειρήσεις και αποτελούν ε, ε, σίγουρα μισθολογική ε, επιβάρυνση όσον αφορά και τη διαμόρφωση των τιμών. Ξέρω δεν είναι ρεαλιστικό ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξουν όλα αυτά και να πούμε θέλουμε να υπάρχει ένα ενιαίο επίπεδο τιμών παντού. Όμως σίγουρα θα ήταν λογικό να πει κανείς αυτές οι εκατοντάδες άτομα δεν είναι οικονομολόγοι, είναι φαρμακευτικά εξειδικευμένα άτομα, είναι ιατροί, φαρμακοποιοί, στις εταιρείε και στις ε, κρατικές αρχές και υπηρεσίες. Και το δυναμικό όλων αυτών για το κόστος, για τα κόστη, το εύρος του κόστους και το δυναμικό εξοικονόμησης ε, μεγάλων ποσών για την κοινωνία μας θα με να το γνωρίζω. Δεν το βρήκα. Ίσως ε, ε, διαβάζοντας μπορεί να μην είναι αυτό άμεσα προσπελάσιμο. Θα ήθελα αυτό σε σχέση με την τεχνολογία να μπορέσει να απαντηθεί διότι θα πρέπει να όταν υπάρχει μια αξιολόγηση να καταλήγουμε σε συμπεράσματα. Δεν είναι δυνατόν, για παράδειγμα, στο, στη Σουηδία να καταλήγουν σε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα από ό,τι στην Ισπανία. Τα πολιτικά συμπεράσματα ίσως μπορεί να είναι διαφορετικά, αλλά για τη μεθοδολογία, για τη μέθοδο, για τους ε, γιατρούς ε, και τους φαρμακοποιούς ε, που για την έρευνα θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξοικονόμηση κόστους. Και τελευταία παρατήρηση στη Γερμανία, στη χώρα μου, στη Γερμανία με βάση τα στοιχεία αυτά τα οποία έχετε, ταξινομείται ως μια χώρα που προσμετρώμενη με το ΑΕΠ της έχει σχετικά υψηλά κόστη φαρμακών. Έχετε κάπου συνυπολογίσει ότι υπάρχει ένα νέο νομοθέτημα εδώ και ένα χρόνο. Ίσως έχει διαδραματίσει ένα ρόλο αυτό. Προσπαθήσαμε να προσαρμόσουμε το επίπεδο, στο ευρωπαϊκό επίπεδο τιμών. Έχετε κάποια στοιχεία ή κάποια συνεργάτες σας για το πώς έχουν διαμορφωθεί αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ. Euh, euh, δεν έχει ε, ζητήσει κάποιο άλλο κάτι. Είχα και εγώ μια ερώτηση εκ μέρου της κυρίας Παρβάνοβα να θέσω. Η κυρία Παρβάνοβα, που λυπάται γιατί δεν μπορεί να είναι μαζί μας σήμερα, θεωρεί ότι η μελέτη αυτή παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον για τις εργασίες μας. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε τις στενού δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσα στην τιμή των φαρμακευτικών προϊόντων και στο θέμα της πρόσβασης στην αγορά της υγείας. Σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιείται για τις μελέτες, η βιβλιογραφία δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολλές ακαδημαϊκές μελέτες, τις οποίες πολλές έχετε κάνει εσείς ο ίδιος κύριε Πρόεδρε. Ένας μεγάλος αριθμός έχει γίνει από τη φαρμακευτική βιομηχανία και πολύ λίγες μελέτες έχουν γίνει από οργανώσεις των ασθενών καταναλωτών πελατών. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια επιπλέον στοιχεία για τις πηγές που χρησιμοποίησατε για τη συγκεκριμένη έρευνα δεν υπάρχουν εργασίες τις οποίες έχουν κάνει ανεξάρτητοι οργανισμοί, οργανώσεις καταναλωτών ή μήπω θεωρήσατε ότι τέτοιες μελέτες δεν ήταν ιδιαίτερα τεκμηριωμένες και δεν τις λάβατε υπόψη σας. Τώρα, σχετικά με την ανάγκη καθορισμού κοινών κατευθυντηρίων γραμμών για την αξιολόγηση των τεχνολογιών της υγείας. Health Technology Assessment θα πρέπει οι διαδικασίες αυτές να περιλαμβάνουν πάρα πολύ μεγάλη βάση τεκμηρίωσης. Λοιπόν, και εσείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχετε να μας κάνετε κάποιες επιμέρους συστάσεις στον τομέα αυτό. Τρίτον, για την σύγκριση και, των διαφορών, και τις διαφορές των τιμών στα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα των γενοσύμων φαρμάκων. Πήρατε υπόψη σας το σύνολο της δυναμικής της αγοράς σε κάθε χώρα που είναι διαφορετική. Η μελέτη δείχνει ότι υπάρχουν πάρα πολύ σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη για τα γενώσιμα σε σχέση με τα πρωτότυπα φάρμακα. Υπάρχουν λοιπόν ειδικά χαρακτηριστικά της αγοράς για τα γενώσιμα που ποικίλει από τη μία χώρα στην άλλη και γι' αυτό εξηγείται και η διαφορά πρόσβασης στην αγορά των προϊόντων αυτών. Τελευταία ερώτηση. Σχετικά με το παράλληλο εμπόριο έχουμε συζητήσει επανειλημμένα. Σας λέτε ότι απαιτείται περισσότερη μελέτη έτσι ώστε να καθοριστεί η επιρροή του φαινομένου αυτού στις τιμές των φαρμάκων. Σε ποιους τομείς οι έρευνες αυτές θα πρέπει να συγκεντρωθούν. Μία ερώτηση για την Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί απαραίτητο να γίνουν αυτές οι έρευνες, θα στηρίξει τις έρευνες αυτές και θα πάρει συγκεκριμένα μέτρα στον τομέα του παραλλήλου εμπορίου. Αυτές είναι οι ερωτήσεις τις οποίες ήθελε να θέσει η κυρία Παρβάνοβα. Η κυρία Μακάβαν έχει στήσει το λόγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη μελέτη η οποία βρήκα ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα με πολλές χρήσιμες πληροφορίες είδαμε πληροφορίες, στοιχεία για κάποια θέματα που είναι δύσκολο να ελέγξει κανείς σχετικά με την πολιτική που ακολουθούν οι ιατροί και τη στάση του κοινού προς τα φάρμακα που είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς. Σε κάποιες ε, ε, χώρες όπως και εδώ πηγαίνει στο γιατρό και ακόμα και για ίσονα προβλήματα υγείας φεύγεις με ολόκληρες σελίδες συνταγογράφησης αν δεν σου δώσει φάρμακα θεωρείται ότι δεν σε εξέτασε προσεκτικά. Ε, θα ήθελα να μάθω αν έχετε κάνει και συγκεκριμένες έρευνες για τα προφίλ για τις ηλικιακέ κατηγορίες, εν πάση περιπτώσει, των διαφορετικών τύπων συνταγογράφησης και σε ποιο βεθμό ε, τα φάρμακα τα... Ε, ξοδεύονται στα τελευταία ένα ή δύο χρόνια της ζωής του ασθενούς γιατί άκουσα ανεκδοτολογικά στοιχεία για πάρα πολλές ποσότητες φαρμάκων σε ηλικιωμένους που δημιουργούν κοκτέιλ τα οποία δεν ξέρουμε πώς λειτουργούν σε επίπεδο αλληλεπιδράσεων αλλά είναι ένα είδος τελευταίας προσπάθειας των γιατρών. Τώρα, προς την Επιτροπή, τι γίνεται με αυτή τη μελέτη. Η μελέτη αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολλά από τα θέματα τα οποία περιλαμβάνει αφορά τις αρμοδιότητες των κρατών μελών, εθνικές αρμοδιότητες. Συζητάτε τα θέματα αυτά σε επίπεδο ομάδων του Συμβουλίου υψηλού επίπεδου. Και τι γίνεται για τις μικρές χώρες. Φαίνεται ότι οι μικρές χώρες υποφέρουν από τον αριθμό των φαρμάκων που τίθεται στην αγορά, που υπάρχουν στην αγορά λόγω του μεγέθους της αγοράς τους. Ε, τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς την κατεύθυνση αυτή. Λοιπόν, πολλά μένει εδώ να γίνουν σε επίπεδο αποφάσεων, ε, σε εθνικό επίπεδο μάλλον αποφάσεων, ισότητας πρόσβασης στα, στα φαρμακευτικά προϊόντα, και ο τρόπος της χρηματοδότησης από πλευράς των ασθενών ε, δείχνει ότι κάποια από τα προϊόντα δεν υπάρχουν σε μια αγορά γιατί το κόστος συγχρηματοδότησης για τον ασθενή είναι πάρα πολύ υψηλό. Λοιπόν, τι γίνεται με αυτές τις ε, μελέτες. Ευχαριστώ. Δεν έχει ζητήσει κανένας άλλος ε, τον λόγο. Θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυρία Λόρα Νίστορ. Καλησπέρα κυρίε και κύριοι. Είμαι η Λόρα Νίστορ. Εκπροσωπώ ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Επιχείρηση. Όπω πολύ σωστά αναφέρθηκε, πρόκειται για αρμοδιότητα των κρατών μελών ο τομέα ε, τη υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα φάρμακα και ιδιαίτερα ε, για τις μικρές χώρες, έχουμε την πλατφόρμα της ε, πρόσβασης ε, στα φαρμακευτικά προϊόντα στην Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτή τη πλατφόρμα έχουμε διάφορε ομάδε εργασία. Για τι μικρέ αγορέ, για παράδειγμα, έχουμε ειδικέ ομάδε εργασία. Όταν συνεδριάζουν τα ενδιαφέρομενα μέρη, συζητούν, προσπαθούν να εντοπίσουν προβλήματα που αντιμετωπίζει η αγορά και να βρουν λύσεις. Πρόκειται λοιπόν για έναν μηχανισμό ανταλλαγής ε, εμπειριών ε, με διεξαγωγή διαφόρων ε, ερευνών ή μελετών μάλλον που μπορούν να βοηθήσουν το έργο αυτών των ομάδων εργασίας. Τώρα, ε, ο σκοπός αυτής της, ε, αυτών των μελετών είναι για να, να τις εξοποιήσουμε εμείς όσο μπορούμε. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και με την ε, μελέτη που έχουμε ενώπιόν μας εδώ. Και γι' αυτό μας ενδιαφέρει εξίσου αυτή η μελέτη με όλες τις άλλες μελέτες που διενεργούνται στον τομέα των φαρμακευτικών προϊόντων αυτή τη στιγμή. Τώρα, σε ό,τι αφορά το παράλληλο εμπόριο, ο συνάδελφος θα μπορούσε να σας πει ενδεχομένω ε, περισσότερα. Γνωρίζετε την ε, θέση του δικαστηρίου, ότι το παράλληλο εμπόριο δηλαδή δεν αντιβαίνει στην συνθήκη. Αυτή είναι λοιπόν η πραγματικότητα, πρέπει να την αποδεχθούμε θα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρον να έχουμε μία έκθεση που θα ποσοτικοποιούσε, αν θέλετε, τα ωφέλη και ε, τα μειονεκτήματα του παράλληλου εμπορίου. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι ε, θα κάνει κάτι επιτροπή σε αυτό το πεδίο. Ευχαριστώ, ελπίζω να απάντησα στις ερωτήσεις σας. Βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε περαιτέρω. Ευχαριστούμε. Ντακμάρ. Με κάθε σεβασμό, όχι, δεν απαντήσατε. Δεν είναι δικό σας το σφάλμα, αλλά εγώ ήμουν μία από αυτούς που πίστευε ότι η φαρμακευτική νομοθεσία είναι στη, καλά κάνει και είναι στη Γενική Διεύθυνση Επιχείρηση. Δεν πρέπει να την πάτε στη Γενική Διεύθυνση Υγεία Καταναλωτών. Όταν όμω την πάτε στη ΣΑΝΚΟ, δεν μπορείτε να αφήσετε ένα τμήμα της οδηγίας για τη διαφάνεια στην Γενική Διεύθυνση Επιχείρηση χωρίς τίποτα άλλο, χωρίς ε, νομική πράξη, χωρίς ε, νομικό πλαίσιο, χωρίς άλλες αρμοδιότητες. Δεν είναι δικό σας το φταίξιμο. Ωστόσο, καλό είναι να, ε, να επιστρέψετε στους ανωτέρους σας και να πείτε να το θέσουν επιτάπητος δεν φταίτε εσεί, αλλά η Γενική Διεύθυνση Επιχείρηση έχει λάξει τι αρμοδιότητέ ε, τη και τώρα ε, μιλάμε για μια σπατάλη χρόνου και πόρων. Και για να είμαι ειλικρινή, ό,τι είπατε δεν μα δίνει κανέν, καμία ένδειξη για τι θα γίνει στο μέλλον. Και δεν φταίτε εσεί, γιατί δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Ε, η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ είναι αυτή που το έχει αναλάβει πλέον. Επομένω, α ε, επαναφέρουμε την τάξη. Ε... Ευχαριστώ. Ο κύριο Καναβός αν μπορείτε να απαντήσετε. Thank you very much, Madam Chair, I'm great. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και τις παρατηρήσεις σας. Όσο μπορώ θα ήθελα ε, να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Το θέμα των φαρμακευτικών προϊόντων είναι ιδιαίτερα περίπλοκο. Είναι αυτονόητο ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλά ενδιαφερόμενα μέρη και δεν το εννοώ αρνητικά. Ε, πολλά διαφορετικά συμφέροντα. Καθώς άκουγα τα ερωτήματά σας, προσπάθησα να τα ταξινομήσω σε κατηγορίες για να απαντήσω κατά τμήματα. Μου φαίνεται ότι υπάρχουν τουλάχιστον τρεις μεγάλες ομάδες. Η πρώτη αφορά το παράλληλο εμπόριο, η δεύτερη την ε, αξιολόγηση, ε, τεχνολογική αξιολόγηση υγείας, η δεύτερη για τις και αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και λόγω της έρευνάς μου. Εγώ θα δώσω τη δική μου οπτική γωνία. Από εκεί πέρα μπορείτε ε, να συναλλαγείτε τα δικά σας συμπεράσματα. Άκουσα το ερώτημα του κυρίου εδώ από την ε, Γερμανία. Ε, για το ενδεχόμενο αποταμιεύσεων από το διασυνοριακό εμπόριο, για την ε, ε, παραποίηση κ.ο.κ. Ας μην ξεχνούμε ότι εδώ έχουμε μία βιομηχανία που αντικατοτρίζει το 1,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Το παράλληλο εμπόριο είναι πολύ μικρό. Ε, συγκριτικά. Οι αποταμιεύσεις είναι ακόμα μικρότερες. Αν δείτε έρευνες που έχουν χρηματοδοτηθεί από ε, τις ενώσεις αυτές ή, την ίδια τη βιομηχανία, αυτές οι αποταμιεύσεις είναι πάρα πολύ μικρές. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα αμελητές. Βεβαίως, ε, ένα τμήμα αυτού του έργου είχε γίνει πριν από 5-6 χρόνια. Πολλά έχουν αλλάξει από τότε. Έχουμε διαφορετικούς τρόπους ε, ε, λειτουργίας πλέον. Τα κράτη-μέλη, για παράδειγμα, απαγορεύουν τις εξαγωγές για λόγους δημόσιας υγείας ή λόγω ελλείψεων. Έχουμε διάφορα τέτοια φαινόμενα. Η δική μου άποψη είναι ότι το θέμα των ενδεχόμενων αποταμιεύσεων, εφόσον ήταν τουλάχιστον ε, μετριοπαθή στο παρελθόν, θα πρέπει να ε, αντισταθμιστούν με τα ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί, μπορούν να προκαλέσουν. Για το παράλληλο εμπόριο μπορούν να, με το παράλληλο εμπόριο μπορούν να υπάρξουν ε, παραποιημένα φάρμακα, ψευδεπίγραφα φάρμακα. Όμως το θέμα αυτό θα υπάρχει πάντα εφόσον ορισμένοι μπορούν ε, να παράξουν ε, φαρμακευτικά προϊόντα ε, στο σπίτι τους. Ίσως είναι πιο εύκολο να υπάρξει δημιουργία ψευδεπίγραφων ή να αποφευχθεί σε ορισμένε περιπτώσει, όπω και να έχει, μπορεί πράγματι να το αυξήσει το παράλληλο εμπόριο ή την ύπαρξη ψευδεπίγραφων φαρμάκων. Για τι πολιτικέ αυτέ, νομίζω από. Ε, ίσως έχουμε υπερβάλει λίγο σε ό,τι αφορά το παράλληλο εμπόριο. Για την ε, τεχνολογική αξιολόγηση στον τομέα της υγείας Βλέπουμε ότι εδώ έχουμε μια μεγάλη δύναμη για την αξιολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων σε όλα τα κρατημέλη. Αυτό που μου προκαλεί εντύπωση και αναφέρεται και στην έκθεση είναι ότι η διαφορά, ε, ότι υπάρχει σημαντική διαφορά ε, στην αξιολόγηση ε, μεταξύ των κρατών μελών, αξιολόγηση των φαρμάκων από κράτος μέλος σε κράτος μέλος ένα κράτο μέλο μπορεί να θεωρεί ικανοποιητικό το φάρμακο, ενώ ένα άλλο όχι και αυτό μπορεί να προκαλέσει διαφορετική διαφορά στην πρόσβαση λόγω ακριβώς ε, αυτής της διαφοράς. Δεν έχουμε συμφωνήσει ακόμα ε, για το πώς ε, αξιολογούμε τις νέες τεχνολογίες. Και αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορούμε να εργαστούμε από κοινού. Πώς αξιολογούμε την καινοτομία δηλαδή και αυτό μπορούμε να το προωθήσουμε περαιτέρω σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να συντονιστούμε περαιτέρω. Υπάρχουν βέβαια ε, ε πρωτοβουλίες, ε, το HTA για παράδειγμα, αλλά είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται και εμείς θέλουμε να την ενισχύσουμε στα επόμενα χρόνια. Η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών βεβαίω και θα βοηθούσε Υπάρχουν κράτη-μέλη βέβαια που ε, λαμβάνουν άλλα κράτη-μέλη ως ε, πρότυπο για τις μελέτες που έχουν γίνει. Τώρα για τα γενώσιμα φάρμακα. Κανεί δεν αμφισβητεί το γεγονός ότι τα ε, φάρμακα είναι πιο φθηνά και μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικές ε, αποταμιεύσεις. Δεν βλέπω όμως κάποια ε, κάποιο πρόβλημα εδώ στο ζήτημα της βιομηχανικής πολιτικής ε, και της ε, προώθησης των γενοσύμων φαρμάκων. Και τα δύο ε, πάνε μια χαρά μαζί μαζί. η διαδικασία παραγωγής δεν, ε, δεν οδηγεί απαραίτητα σε αύξηση της αποσχόλησης γιατί είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία πλέον, αλλά σε μια, στην αύξηση της έρευνας η βιομηχανία που βασίζεται στην έρευνα ε, συμβάλλει ιδιαίτερα στην έρευνα και την ανάπτυξη, αλλά και στην απασχόληση. Δεν βλέπω λοιπόν κάποιο πρόβλημα εδώ. Ούτε υπάρχει ε, διαφορά ανάμεσα στην ε, προώθηση της χρήσης ενός οικονομικά αποδοτικού προϊόντος και στην εξοικονόμηση πόρων για την διοχέτευσή τους κάπου αλλού. τι μπορούμε να πιστέψουμε και τι όχι. Υπάρχουν ε, πολλά δεδομένα και πληροφορίες ε, για την επίδοση, για τις επιδόσεις ε, της βιομηχανίας ή μεμονωμένων πολιτικών. Αλλά χρειαζόμαστε μία πραγματική αξιολόγηση. Τώρα, το αν ε, η έρευνα και η ανάπτυξη είναι 15%, αν αυτό είναι μικρό, χαμηλό ή υψηλό ποσοστό. Για μένα είναι αρκετά σημαντικό αυτό το ποσοστό του συνολικού δηλαδή φαρμακευτικού κόστους. Ας μην ξεχνούμε όμως ότι κατά πάσα πιθανότητα είναι, είναι ε, μεγαλύτερο γιατί εμείς ως φορολογούμενοι άμεσα ή έμεσα συμβάλλουμε στις εθνικές ε, ε, πολιτικές στην έρευνα και ανάπτυξη. Δεν είναι δηλαδή μόνο η φαρμακευτική βιομηχανία που επενδύει στην έρευνα και στην ανάπτυξη αλλά και οι ευρωπαίοι φορολογούμενοι είτε σε εθνικό επίπεδο είτε και σε ευρωπαϊκό. Αυτό απαντά και στο ερώτημα για τα ε, price funds, τα κονδύλια ε, κοστολόγησης. Δηλαδή πώς θα ε, προωθήσουμε την καινοτομία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εγώ δεν είμαι κατά αυτής της ιδέας, θα μπορούσα να τη στηρίξω, αλλά θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πιο ανοιχτό ε, μοντέλο ή πρότυπο καινοτομίας. Τα κράτη-μέλη αλλά και η βιομηχανία το αναγνωρίζει αυτό, λένε και περισσότερο. Κάτι άλλο που αναφέρθηκε προηγουμένως για το ποιος ε, κερδίζει εδώ τις εξελίξεις ε, στα μεμονωμένα κράτη-μέλη είναι ένας τομέας πολιτικής με ιδιαίτερη δυναμική. Γιατί με το που δημοσιεύθηκε η έρευνα αυτή πριν από μερικού μήνε είναι ήδη παροχημένη. Γιατί αναφέρεται σε στοιχεία ε, τριών ετών. Είναι ένας τομέας που αλλάζει συνεχώς. Είτε μιλάμε για τις εξελίξεις ό,τι αφορά τι τιμέ, είτε για τι αποταμιεύσει από τα γενώσιμα φάρμακα και ούτω καθεξής. Τι να πιστέψουμε και τι όχι μπορούμε να πιστέψουμε τα ε, στοιχεία που μας ε, ε, παρέχονται, εφόσον αυτά παρέχονται με τον κατάλληλο και ενδεδειγμένο τρόπο, όταν ακούγονται όλες οι διαφορετικές φωνές, γιατί υπάρχουν διαφορετικές φωνές και απόψεις. Αυτές λοιπόν θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται επαρκώς και σωστά. Και από εκεί πέρα οι ευρωβουλευτές μπορούν να αντιλήσουν τα δικά τους συμπεράσματα για το τι συμβαίνει. Η δυναμική μεταβάλλεται συνεχώς. στα μεμονωμένα κατημέλη. Βεβαίως και υπάρχουν ζητήματα ε, κοστολόγηση, αλλά υπάρχουν και ζητήματα όγκου που αφορούν μεγάλες αλλά και μικρές χώρες. Στο τελευταίο σημείο επανέρχομαι στο διασυνοριακό εμπόριο ε, για το πού θα πρέπει να εστιάσει η έρευνα ίσως αν υπάρχει ανάγκη, αλλά για να κατανοήσουμε απλώς ε, το τι συμβαίνει ή τα ωφέλη και τα μειονεκτήματα. Έχουν γίνει ε, μελέτες σε αυτό το τομέα από μένα αλλά και από άλλους. Επειδή όμως η δυναμική αυτή, η δυναμική συνεχώς, καλύτερα είναι να εστιάσουμε κάπου αλλού. Η Λόρα Νίστον από την Επιτροπή ανέφερε ορισμένα πράγματα. Τώρα η Επιτροπή, αν πρόκειται για την Digin Σάνκο ή για την ε, Γενική Διεύθυνση Επιχείρηση, ε, εργάζονται σκληρά αν και κοιτάξετε την κατάσταση πριν από 10-15 χρόνια, όταν κάτι μέλη ούτε καν συζητούσαν το ενδεχόμενο ανταλλαγή ε, βέλτιστων πρακτικών, ε, μπορώ πλέον να σας πω ότι τα κράτη-μέλη ε, συζητούν ε, και ανταλλάσσουν τέτοιες εμπειρίες. και να ανταλλάξουν απόψεις για το αν κάτι λειτουργεί στην επικράτειά τους είτε όχι. Η Επιτροπή λοιπόν έχει δραματίσει ένα ρόλο σε αυτό, χωρίς βέβαια να θέλω να ε, υποβαθμίσω αυτό που ε, μας είπατε εσείς. Κύριε Πρόεδρε, πολλά αναφέρθηκαν. Ελπίζω να απάντησα ε, σε ορισμένα από αυτά τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Σε ευχαριστώ για τις απαντήσεις σου, τις πληρέστατες, τις ερωτήσεις που θέσαμε. Ευχαριστούμε για την ποιότητα της έκθεσης και για αυτή την οπτική γωνία που μας προσέφερε σήμερα για ένα σημαντικό θέμα. Προκαλέσατε το ενδιαφέρον των συναδέλφων. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ε, λεπτομέρειες τις οποίες έκανε, αν και εδώ θα συμφωνήσω με την κυρία Ροτ Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο, ε, πρόεδρος από εδώ και πέρα θα συνεχίσει ο κύριος Σλίτερ, του δίνω το λόγο. Του δίνω την προεδρία μάλλον πρώτα.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 Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Είναι η παρουσίαση του ECDC για τις υπατήτηδες Β και Γ. Έχω μαζί μας τον κύριο Σπρίγκερ, ο οποίος είναι Γενικός Διευθυντής Ελπίζω να μπορέσετε να επιστρέψετε. Από ό,τι φαίνεται ότι ε, θα φτάσουν στην Ανατολική Σουηδία το απόγευμα, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε πάρα πολλές διαφορές σε ορισμένες χώρες, έχουμε αυξημένα ε, κρούσματα, σε άλλες λιγότερο. Ευχαριστώ. Και εγώ ελπίζω να επιστρέψω στο Κόλμη, λέει ο κ. Σπρέγκερ. Ξέρω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται ιδιαίτερα στην υπατήτηδα Β και στην υπατήτηδα Γ και αυτό με χαροποιεί. Παρατήρησε επίσης ότι υπάρχει μια δήλωση ήδη από το 2007 και ζητάτε ήδη από το 2007 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει συστάσεις σχετικά με τον έλεγχο για την ασθένεια αυτή. Καθολικού τύπου έλεγχο. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει να ληφθούν ορισμένα μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι οι πατήτηδες Β και Γ ε, υπάρχει υποχρέωση να δηλώνονται σε επίπεδο ECDC και σε διεθνές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε λοιπόν πολλά στοιχεία. Το 2007 δώσαμε μια πρώτη εικόνα της κατάστασης σχετικά με τις υπατήτηδες αυτές. Η εικόνα αυτή αφορούσε την περίοδο 1995 με 2004, 10 χρόνια. Τώρα όμως είμαστε σε θέση να δίνουμε ετήσια στοιχεία. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι σοβαροί περιορισμοί. Πάντα τίθεται το θέμα. Αν βλέπει κανείς μια αύξηση, αυτή η αύξηση τι μπορεί να σημαίνει. Σημαίνει ότι οι ιατροί δίνουν περισσότερη προσοχή στη συγκεκριμένη ασθένεια και την ελέγχουν περισσότερο. Υπάρχει πράγματι αύξηση των κρουσμάτων. Μια αύξηση λοιπόν στον αριθμό των κρουσμάτων είναι πάρα πολύ δύσκολο να ερμηνευθεί. Συγκεντρώσαμε πάρα πολλούς εμπειρογνώμονες και αρχίσαμε να συζητάμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αξιολογήσουμε το πραγματικό βάρος της ασθένειας αυτής και να δούμε αν μπορούμε στη συνέχεια να διαμορφώσουμε κάποιες επιλογές. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει το πρόβλημα, χιλιάδες πολιτών μολύνονται από τη συγκεκριμένη ασθένεια και πάρα πολλοί οδηγούν σε κυρώσεις του ύπατος, οδηγούνται σε κυρώσεις του ύπατος και κάποιοι σε υπατικούς καρκίνους δεν κατανέμεται ισότιμα το βάρος της ασθένειας αυτής. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές και αυτό είναι κάτι το οποίο σας ενδιαφέρει. Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη και στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Και αυτό φαίνεται από την έκθεσή μας. Σαν παράδειγμα, η πατήτηδα γάμα συγκεντρώνεται βαρύτατα ανάμεσα στους ενέσιμους χρήστες ναρκωτικών, και οι οποίοι εκτίθενται σε υψηλό επίπεδο κινδύνου και για την Β και για την Γ. Θα ήθελα να κάνω τώρα ορισμένα σχόλια για το τι ακριβώς κάνουμε σχετικά με τις ασθένειες αυτές. Η υπατήτηδα Β μπορεί να προληφθεί μέσω της ε, σωστής ε, μεθόδου εμβολιασμού που είναι διαθέσιμη εδώ και 20 χρόνια, είναι επιτυχεστάτη είναι πολύ αποτελεσματική και τα ποσοστά έπεσαν από 10 περιπτώσεις υπατήτηδας Β σε 100.000 πολίτες το 1994 σε μία. Έχει μειωθεί κατά 10 ε, φορές δηλαδή η ε, ασθένεια αυτή. Βέβαια ε, στους ναρκωμανείς που είναι μία από τις υψηλές ομάδες κινδύνου και για τη Β και για τη Γ υπάρχει αύξηση. Προσπαθήσαμε λοιπόν μαζί με το Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και των Εξαρτήσεων από Ουσίες, αναπτύξαμε ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για το πώς μπορούμε να αναλάβουμε κάποιες δράσεις στον συγκεκριμένο τομέα. Αν εντοπιστούν αρκετά ενωρίς, πολλοί που υποφέρουν από υπατήτηδα γάμα μπορεί να θεραπευθούν. Αυτοί μπορούν να, να, να τους φροντίσει κανείς φαρμακευτικά αυτούς που υποφέρουν από τη β αλλά το πρόβλημα είναι ο έλεγχος. Ο σωστός έλεγχος, ο ιατρικός, απαιτεί πάρα, ε, πολλά χρήματα και το θέμα είναι αν ε, αξίζει τον κόπο να ξοδέψει κανείς τόσα χρήματα. Γιατί ε, αν εντοπιστούν κρούσματα θα πρέπει να παρέχεται θεραπεία και η θεραπεία κοστίζει. Γι' αυτό ακριβώς το ECDC προσπαθεί να αναπτύξει ένα πρότυπο για την αξιολόγηση των μεθόδων ελέγχου είναι ένα, μια εργαλειοθήκη για την υπολογισμό, για τη σχέση κόστους αποτελέσματος σε εθνικό επίπεδο. Θα καταστήσουμε τα αποτελέσματα αυτά διαθέσιμα στις αρχές του επομένου έτους και θα θέλαμε να προσκαλέσουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τα μέσα αυτά και να λάβουν υπόψη τους τη δική τους κατάσταση και να δουν αν τα μέσα αυτά θα τους οδηγήσουν στο να ξεκινήσουν προγράμματα ελέγχου του πληθυσμού. Το 2012 και πέραν θα έχουμε ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων στα κράτη-μέλη για να αναπτύξουμε ένα πλαίσιο πρόληψης και ελέγχου της υπατήτηδας Β και Γ. Ένα θέμα το οποίο ήδη έχει εντοπιστεί σαν προτεραιότητα είναι η πρόληψη η μετάδοση από μητέρα σε παιδί τη υπατήτηδα Β. Αυτό μπορεί να γίνει ευθυνότατα και απλά, εφόσον γνωρίζουμε βέβαια ότι η μητέρα είναι μολυσμένη. Εξεπλάγει από ότι έμαθα ότι υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη τα οποία δεν ε, ελέγχουν τις εγγύου γυναίκες για την υπατήτηδα Β συστηματικά. Αυτό ελπίζω να αλλάξει. Είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να συνεργαστούμε για να αλλάξει. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Okay, thank you. Well, uh, I'll start with, uh, or maybe actually, it, I, I heard that Laszlo Benze is. Άκουσα ότι Laszlo Λάσλο Μπέντσα είναι εδώ από το Συμβούλιο. Πώς θέλετε να πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. a tanács részéről a magyar elnökség alatt a népegészség. Όσον αφορά την ίδια την Προεδρία, εγώ είμαι επικεφαλή τη ομάδα εργασία για την δημόσια υγεία. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που μπορώ να παραστώ και η εισήγηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα για μένα, πρέπει να πω. Τώρα, θα ήθελα στη συνέχεια από πλευρά τη ομάδα Εργασίας για την Δημόσια Υγεία να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Προσέξτε, η Ουγγρική Προεδρία έχει συνειδητοποιήσει σαφώς το γεγονός ότι έχει συνδέονται πολύ σοβαρά προβλήματα με την υπατήτη Β και Γ και το γνωρίζουμε αυτό και εκτιμούμε ιδιαίτερα τις δραστηριότητες ε, της ECDC ε, του Ευρωπαϊκού Κέντρου και γνωρίζουμε ότι πολλά περισσότερα ακόμα πρέπει να πράξουμε ώστε τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν και να επιληθούν όσον αφορά το πρόγραμμα της ίδιας της Ουγγρικής Προεδρίας γνωρίζετε ότι οι δυνατότητες μας είναι περιορισμένες βέβαια έπρεπε κάποιες προτεραιότητες να θεσπίσουμε, να καταρτήσουμε, επί των οποίων θα επικεντρωνόμαστε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας και έτσι έχουμε τέσσερις τομείς που ταυτοποιήσαμε, εντοπίσαμε όπου συμπεράσματα του, της Προεδρίας θα θέλαμε να εγκριθούν και θα θέλαμε από πλευράς μας το Ειδικό Συμβούλιο, να, το Συμβούλιο να μπορέσει να εγκρίνει τέσσερις, τέσσερα, τέσσερις προτάσεις από πλευράς της Ουγγρικής Προεδρίας για αυτά. Επιλέξαμε μια διαφορετική κάπως προσέγγιση από αυτά τα οποία προαναφέρθηκαν, διότι η δική μας προσέγγιση είναι εξειδικευμένη όσον αφορά την, την, τις ασθένειες και τις επιπτώσεις τους ε, στην δημόσια υγεία. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό των ασθενειών και της καταπολέμησής τους ε, για τη δημόσια υγεία επικεντρωνόμαστε τα εμβόλια κατά των, ε, κατά των ασθενειών αυτών, ιδιαίτερα εμβολιασμούς νέων ανηλίκων παιδιών. Σε αυτά επικεντρωνόμαστε, σκεπτόμαστε ότι οι προστατευτικοί αυτοί εμβολιασμοί κατά την παιδική ηλικία ε, αποτελούν μια, μπορούν να αποτελέσουν μια μεγάλη πρόσθετη αξία για την Ευρώπη. Εξάλλου πιστεύουμε ότι η Ουγγαρία όσον αφορά αυτό το ζήτημα έχει θετικές ε, εμπειρίες ε, και βιώματα επ' αυτών και αυτοί οι δύο λόγοι είναι εκείνοι που μας έκαναν να αποφασίσουμε να πορευτούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε αυτές λοιπόν τις αποφάσεις που προτείνουμε να εγκριθούν από το Συμβούλιο θέλουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να ζητήσουμε μέσα στο πλαίσιο των εμβολιασμών των εμβολίων και εμβολιασμών να δραστηριοποιηθούν, δραστηριοποιηθούν περισσότερο. Ζητούμε να ενταθεί η εργασία, να ενταθεί η έρευνα, οι δραστηριότητες γύρω από την έρευνα και θεωρούμε επίσης ότι τα αποτελέσματα σε αυτό τον τομέα μπορούν να συνεισφέρουν και να είναι πολύ θετικά και έτσι καλύτερα να καταπολεμήσουμε την υπατήτηδα Β και Γ οι Β και Γ υπατήτηδες ε, δεν έχουν εγγραφεί συγκεκριμένα εξειδικευμένα στη μέρησια διάταξη του Συμβουλίου και με τις προτάσεις αυτές, αλλά έμεσα μπορούμε να συνεισφέρουμε ώστε η καταπολέμηση αυτών των ασθενειών να ενταχθεί στα πλαίσια αυτά. Σας ευχαριστώ, αναμένω προσδοκώ σε ερωτήσεις σας. Να δώσω το λόγο τώρα στα μέλη και μετά δώσω το λόγο βέβαια και στην Επιτροπή για να απαντήσει. Διάβασα και πάλι στην ημερήσια διάταξη αναφέρεται τρέχουσες πρωτοβουλίες για την καταπολέμηση της υπατήτηδας Β και Γ και περαιτέρω προτάσεις. Περαιτέρω προτάσεις. Σε αυτές τις περαιτέρω προτάσεις θα ήθελα να αναφερθώ στην παρέμβασή μου. Ένας από, να το πω, από τους κυριότερους λόγους για τη δημιουργία και την συγκρότηση του ECDC ήταν το θέμα της καταπολέμησης των μεταδιδόμενων μολυσματικών ασθενειών. Αυτή τη στιγμή έχουμε, πώς να το πω, μια, ένα μεγαλύτερο κύμα μιας ε, τέτοιας ε, ε, προσβολής των χωρών μας στη Γερμανία με το AIDS και, το, και τους ιούς αυτούς που οδηγούν σε πραγματικά πολύ σοβαρές καταστάσεις όπως στην Γερμανία. Ένας αυξημένος αριθμός ατόμων βρίσκονται σε, σε εντατική, στους εντατικούς Ερώτηση, τι κάνει σε σχέση με το ECDC, υπάρχουν ε, ειδικέ task force που έχουν ε, συγκροτηθεί, υπάρχουν δυνατότητες ε, παροχής βοήθειας ώστε τα αίτια αυτών των, αυτών των μολύνσεων να αναζητηθούν και να διαρευνηθούν και για την παραμονή των ασθενών αυτών ε, να έχει ληφθεί υπόψη ότι για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει ο κίνδυνος μετάδοσης, μόλυνσης. Είναι σημαντικά αυτά τα θέματα. Αντιμετωπίζουμε εδώ και πολλά χρόνια το ζήτημα της υπατήτας Β και Γ. Αλλά τώρα όταν έχουμε μία ασθένεια που έχει ε, παρατηρηθεί εδώ και μερικές ημέρες για παράδειγμα, ίσως θα μπορούσε το ECDC να εντείνει την ε, σημασία των προσπαθειών του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήματα. Πρώτον, να ευχαριστήσω τον συνάδελφο για την παρουσίαση για τον ECDC. Όπως είπε και Ντάγμα, είναι ένας πολύ καλός οργανισμός, αν θέλετε, για τη συλλογή δεδομένων και πάντα με ενημερώνει όταν υπάρχει ένα πρόβλημα. Ε, ακούσαμε και τον Μάρκ, είπε ότι ήδη καταβάλει προσπάθειες για το ζήτημα της μετανάστευσης ε, που ε, πλήττει ορισμένα σε επίπεδο διάδοσης ασθενειών. Δύο ερωτήματα λοιπόν. Πρώτον είπατε ότι τα κράτη-μέλη έχουν διαφορές στην υπατήτηδα Β και Γ. Αυτό γιατί συμβαίνει. Επειδή υπάρχει διαφορετικό επίπεδο ευαισθητοποίηση στα κράτη-μέλη, επειδή υπάρχουν περισσότερε ευάλωτε ομάδε, ε, ε, ε, είναι πολιτισμικό το γεγονό. Σε τι οφείλονται αυτέ οι διαφορέ, λοιπόν. Ε, Επίσης αυτό εμφανίζεται και σε ε, διασυνοριακό επίπεδο. Μετά για τα προγράμματα ανείχνευσης, screening είναι ευαίσθητο ζήτημα γιατί ε, βεβαίως ανακύπτουν ζητήματα όπως αν θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό ή ε, προαιρετικό, αν θα ασφαλίζεται και τι γίνεται όταν μάθεις στο τέλος τι συμβαίνει. Γενικά συμφωνείτε ότι είστε υπέρ ενός προγράμματος ανείχνευσης ε, ενάντια στις μολυσματικές ασθένειες. Αν μπορείτε να μας απαντήσετε. Ευχαριστώ. Ελιζαμπέτα Λουκασεύσκα. E, e, e, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μας ε, δώσε απευθύνατε. Θέλω να ευχαριστήσω για τις πληροφορίες. Θα ήθελα να γνωρίζω, να μου πείτε, Ήθελα σε σχέση με την υπατήτητα Β σε σχέση συγκεκριμένες χώρες να μάθω τα εξή. Βλέπει κανείς συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ των χωρών αυτών. Σωστό, αναφέρατε ότι η καταπολέμηση της ε, υπατήτηδας όσον αφορά τις δραστηριότητες, ε, τις συγκεκριμένες δραστηριότητες έγκυται το screening στις εξετάσεις όσο το δυνατόν νωρίτερα. Είναι όμως μια δαπανηρή μέθοδος και δεν γίνεται συχνά χρήση αυτής της μεθόδου. Πιστεύω ότι σε πολλές ασθένειες όσον αφορά το φθηνότερο τρόπο η προφύλαξη, η πρόληψη είναι η καλύτερη οδός. Δεν έχετε πει όμως, δεν αναφέρετε τίποτα σε σχέση με αυτό και σε σχέση με τον πληθυσμό και τα προφυλακτικά μέτρα πρόνοιας, προληπτικά. Τι γίνεται, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Καρίν Κάνταμας. Ευχαριστώ και μετά θα ήθελα σε σχέση με τις ε, παρατηρήσεις ε, να αναφερθώ και από την Προεδρία του Συμβουλίου οι εμβολιασμοί των παιδιών αναφέρθηκαν ως πρωτοβουλία ώστε να ανοσοποιηθούν τα παιδιά σε κάποια κράτη-μέλη έχουμε τέτοιου είδους ε, προγράμματα ως ε, μέτρα υποσύσταση που πρέπει να ακολουθηθούν. Στην Ευρώπη, Ευρώπη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε το πρόβλημα αυτό και ερώτηση είναι ποια προγράμματα και σχέδια υπάρχουν από, τη, από πλευρά σας. Υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, μήπως ε, φταίνε τα εμβόλια ή φταίει η κόποση ή μη ιδιαίτερη προθυμία για εμβολιασμού. Τι συμβαίνει σε αυτό το πεδίο. Ευχαριστώ. Thank you. I have no more members. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητά κάποιο άλλο το λόγο. Θα δώσω λοιπόν πρώτα το λόγο στην Επιτροπή και μετά στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψη και Ελέγχου Νόσων. Σαφρανή, νομίζω. Α, ah, John Ryan. Καλησπέρα. Αρχικά σας ευχαριστώ που το συζητούμε αυτό το θέμα σήμερα. Είναι σημαντικό να συζητείτε ανατακτά χρονικά διαστήματα στο βήμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί ε, βεβαίως και ε, ελκύει μεγαλύτερη, περισσότερο ενδιαφέρον, αν θέλετε, εδώ. Υπήρξαν πρωτοβουλίες και στο παρελθόν και το 2007, αλλά και από τον ΠΟΗ για το ίδιο θέμα. Είναι πολύ χρήσιμο λοιπόν ε, να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον ε, για τη συγκεκριμένη αυτή ασθένεια. Από το 2000 και μετά η Επιτροπή έχει αναγνωρίσει την ανάγκη ε, ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών ενάντια σε αυτόν τον ιό Μπορώ να σας πω συγκεκριμένα ότι η νομοθεσία που έχουμε για την ε, επιτήρηση των μεταδοτικών ασθενειών έχει καλύψει την υπατήτηδα Β και Γ, υποχρεώνοντας τα κράτη-μέλη να, ε, να ε, υποβάλουν εκθέσεις ε, ανατακτά χρονικά διαστήματα για τα κρούσματα υπατήτηδας Β και Γ. Επιπλέον, θα ήθελα να πω ότι το, Ευρωπαϊ... το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υγεία έχει χρηματοδοτήσει και θα εξακολουθήσει να χρηματοδοτεί ε, μια σειρά προγραμμάτων που στοχεύουν συγκεκριμένα στην υπατήτηδα. Ε, θα χρηματοδοτήσουν για παράδειγμα την, ε, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, την κατάρτιση των, του προσωπικού υγειονομικής περιθάλψης, ε, ανάπτυξη των προληπτικών μέτρων για την υπατήτητα Β και Γ και την ενημέρωση συγκεκριμένων ομάδων, ε, πληθυσμιακών ομάδων. Έχουμε ήδη ακούσει τις συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Ένα παράδειγμα είναι ένα ε, πρόγραμμα συσχετισμού που μπορεί να αναπτύξει προσέγγιση των αιματογενώς μεταδιδόμενων νόσων για τους ναρκωμανείς συγκεκριμένα προγράμματα για την πρόληψη στις φυλακές και ένα τρίτο πρόγραμμα για την πρόσβαση στην περίθαλψη για ε, αλκοολικούς και ναρκωμανείς. Τώρα στην Επιτροπή συζητούμε ένα επιπλέον ε, πρόγραμμα για φέτος για την ανείχνευση της υπατήτηδας και έχουμε συνάντηση με τους ε, συντονιστές του προγράμματος. Ο στόχος ε, εδώ είναι να αναπτύξουμε κοινέ προσεγγίσεις για τα προγράμματα ανείχνευσης, ε, να βοηθήσουμε τις προμήθειες και συγκεκριμένα να εστιάσουμε στις εθνωτικές μειονότητες. Βεβαίως πολλά μένουν ακόμα να γίνουν η πατήτητα Β και Γ ε, εξακολουθούν να αποτελούν ε, ε, κινδύνους για τη δημόσια υγεία και αναγνωρίζουμε την ανάγκη υπέρξης περαιτέρω πρωτοβουλειών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό και ζητήσαμε από τον ECDC το 2009 να διενεργήσει μελέτες για την υπατήτητα Β και Γ. Στόχος ήταν να συλλέξουμε ανεξάρτητες και άρτιες επιστημονικές ενδείξεις για το βάρος της ασθένειας, αλλά και για την αποτελεσματικότητα ενδεχόμενων μέτρων πρόληψης και ελέγχου. Το 2010 το ECDC εξέδωσε μια πρώτη σειρά μελετών ε, που τόνισε την ετερογένεια του φαινομένου στο Ευρωπαϊκό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον περισμένο αριθμό πληροφοριών ε, για την προστιθέμενη αξία της ανείχνευσης. Έχουμε περαιτέρω ε, δραστηριότητες σε πλαίσιο ECDC για να καλύψουμε αυτά τα κενά. Κατανοούμε ότι αυτά τα μέτρα ε, και όλες αυτές τις προσπάθειες απαιτούν χρόνο. Ωστόσο, είναι σημαντικό τα μέτρα που προτείνουμε στα κράτη-μέλη βασίζονται σε δεδομένες αποδείξεις. Και θα εξαρτηθεί και από την ε, δυνατότητα του ECDC να μας παράσχει αυτά τα δεδομένα. Στην Επιτροπή συνεχίζουμε λοιπόν το έργο μας για την πρόληψη και την θεραπεία της επατήτητας Β και Γ βάσει και των ε, ε, διατάξεων του ψηφίσματος της Ολομέλειας του ΠΟΗ και θα προσπαθήσουμε αυτό να το κάνουμε μέχρι τα τέλη του χρόνου. Να βελτιώσουμε δηλαδή τα επίπεδα επιτήρηση ε, για την υπατήτητα Β και Γ σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα μα επιτρέψει να συγκρίνουμε μεγαλύτερη άνεση τα δεδομένα ε, για να εντοπίσουμε το βάρο τη ασθένεια. Ε, Βεβαίω και συνεχίζουμε να χρηματοδοτούμε προγράμματα υγειονομικά για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών, την σύνταξη κατευθυντήριων γραμμών, αλλά και εξαρτή ενημέρωση προ συγκεκριμένε πληθυσμιακέ ομάδε. Όπω είπε και ο πρόεδρο ε, του Συμβουλίου, τη Ομάδα Εργασία του Συμβουλίου, ε, το Συμβούλιο θα υιοθετήσει στι 6 Ιουνίου ε, συμπεράσματα του Συμβουλίου για, την, για τον εμβολιασμό των παιδιών. Και αυτό βεβαίω και θα συμβάλλει στην προστασία του κοινού η Επιτροπή στη συνέχεια θα αναλύσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου μετά την υιοθέτησή του για να δούμε πώς μπορούμε να το συνδέσουμε αυτό το θέμα με το θέμα της υπατήτηδα, με την πρόληψη και τον έλεγχο. Και απαντώντα ε, στην συνάδελφο Ντάγμα Ρορ Μπέρεντ, οι γερμανικές αρχές μας έχουν ενημερώσει για τα κρούσματα αυτά με το, ε, με το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Και καλέσαμε ε, τον ECDC να κάνει μια αξιολόγηση κινδύνου. Και όταν γίνει αυτό, όταν τη λάβουμε αυτή την αξιολόγηση, θα ε, συναντηθούμε με τα κράτη-μέλη για να εντοπίσουμε συγκεκριμένα μέτρα που μπορούν να ληφθούν. Και βεβαίως και τις αρχές επιστηστικής ασφάλειας. Ευχαριστώ. Βεβαίως ε, είμαι περίεργος να μάθω πόσο χρόνο θα πάρει μια τέτοια αξιολόγηση κινδύνου. Ε, ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς την Ουγγρική Προεδρία γιατί έχει δώσει πάρα πολύ προσοχή στην, στον εμβολιασμό των παιδιών. Οργανώσαμε από κοινού μια διάσκεψη εμπειρογνωμόνων και είμαστε ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα ιδιαίτερα. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον εμβολιασμό των παιδιών και στην ε, αύξηση των ε, μολύνσεων των παιδιών σχετικά με την, ε, με την υπατήτηδα σε καθημερινή βάση με την γερμανική υπηρεσία, όποτε είμαι στο γραφείο παίρνω μέρος σε μια συνάντηση που γίνεται ηλεκτρονικά και η ηλεκτρονική απάντηση επίσημη είναι ότι θα δραστηριοποιείται το σύστημα μετά από αίτημα του κράτους μέλους. Παρακολουθούμε όμως και εξωτερικά μηνύματα, τα μέσα ενημέρωσης και τα λοιπά, ακόμα και τα Σαββατοκύριακα βλέπουμε τις ανεπίσημες έρευνές μας, αλλά δεν μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε μετά από επίσημο αίτημα μόνο. Χθε ας πούμε το μήνυμα είναι ότι υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο αφορούσε τη Γερμανία, εφόσον υπάρχει μόνο σε μία χώρα μέλος, το ECDC θα ζητήσει τη γνώμη φυσικά του κράτους μέλους για να παρέμβει. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια υπηρεσία για γρήγορη αξιολόγηση του κινδύνου. Μπορούμε να παράσχουμε μια τέτοια μελέτη σε επίπεδο 48 ώρων. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα πρόσφατα. Υπήρξαν περιπτώσεις ε, κάποιων, ε, uh, κάποιων μορφών πυρετού μολυσματικού προσπαθήσαμε να το ελέγξουμε εκεί όπου είχαν συγκεντρωθεί τα κρούσματα σε, σε τουριστικές περιοχές και εκεί υπάρχει θέμα φυσικά και με τα προβλήματα υγιεινής των ε, ξενοδοχείων. Για την κυρία Γιανακουδάκη μας είπε ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι πληθυσμού αυτό αφορά επίσης και προβλήματα όπως ε, τους ε, χρήστες ναρκωτικών όπως είπα, όπως ε, τους εξαρτημένους από το αλκοόλ. Είναι πάρα πολύ εύκολο να πει κανείς να βγει να πει ότι εντάξει ας ελέγξουμε όλο τον κόσμο. Αλλά η ασθένεια αυτή συγκεντρώνεται ιδιαίτερα σε πληθυσμού όπω οι χρήστε των ναρκωτικών, οπότε τι νόημα έχει να ελέγξει το σύνολο του πληθυσμού. Εγώ είμαι υπέρ μια επιλεκτική αντιμετώπιση και να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα που έχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν είμαι γενικά υπέρ των προγραμμάτων ελέγχου του πληθυσμού. Πρέπει κατά περίπτωση να δούμε αν αυτό αξίζει και αν αξίζει να επενδύσουμε στον έλεγχο και ποιε είναι οι ομάδε που θα πρέπει να ελεγχθούν. και μόνο εφόσον υπάρχει δυνατότητα θεραπείας της ασθένειας, γιατί δεν έχει νόημα να διαπιστώνει κανείς την ύπαρξη μιας ασθένειας σε ένα ασθενή και να μην είναι σε θέση να παράσχει την θεραπεία. Και για το, για το AIDS επίσης εμένουμε φυσικά στο θέμα του ελέγχου. Εκεί υπάρχει θέμα σε σχέση με την παροχή σωστής θεραπείας σε όλα τα κρατη για την ερώτηση Κάλεμπαχ. Ξέρετε ότι υπάρχει πρόβλημα με την παροτίτιδα στην Ευρώπη. Oh, um, Ήταν ασθένεια κυρίως παιδική, αλλά τώρα βλέπουμε να υπάρχουν προβλήματα. Το 30 περίπου της 100 των περιπτώσεων χρήζουν ε, θεραπεία σε νοσοκομιακό χώρο σε ενηλίκους και νομίζω ότι εκεί ε, μιας και έχουμε την δυνατότητα εμβολιασμού θα ήταν καλό. Είναι κρίμα γιατί εξάγουμε εμεί ουσιαστικά αυτή την ασθένεια στον υπόλοιπο κόσμο και δεν την ελέγχουμε. Δεν είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι θέμα κρατών μελών. Έχουμε όμως ήδη ε, σημάνει τον κόδωνα ε, του κινδύνου. Λοιπόν, ζητάμε να υπάρξει συντονισμένη αντίδραση. Η καταπολέμηση ε, της ε, παροτίτιδας δεν αρκεί από μόνη της. Θα πρέπει να πείσουμε και τους γιατρούς να στρέψουν την προσοχή τους, ε, τα κοινωνικά μέσα και επίσης να προειδοποιήσουμε και τους γονείς και να τους πείσουμε ότι η ασθένεια αυτή είναι πολύ σοβαρή και πρέπει να εμβολιαστεί ο πληθυσμός εναντίον αυτής της ασθένειας. Είναι ευθυνός και ασφαλής ο εμβολιασμός. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Σας εύχομαι καλό ταξίδι στη Στοκόλμη. Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι το γλυκό θέμα των μελισσών. Ξέρουμε βέβαια δεν είναι και τόσο γλυκό. Έχουν υπάρξει πολλά προβλήματα υγείας. Δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρόβλημα με τον πληθυσμό των μελισσών, αλλά υπάρχει μείωση ε, αυτού του είδους των εντόμων, που είναι η συγχύτριά μας. Η Τζούλι Γκέρλινγκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα κάνω μια πολύ σύντομη εισαγωγή. Θα ξεκινήσω με αυτά τα οποία λέγουν προκαταρκτικά αυτοί οι οποίοι δίνουν τις νομοδοτήσεις ότι υπάρχει ένα θέμα συλλογής πληροφοριών Πολλές από τις πληροφορίες δεν είναι πάρα πολύ γνωστές. Στην ουσία αυτά τα οποία θα πω είναι περισσότερο θέματα προσυζήτηση παρά στοιχεία. Να πω ότι προσπάθησα να αναφερθώ σε πολλά θέματα, σε όλα τα θέματα, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα γύρω από τις μέλωσες. Πολλά από αυτά θα πρέπει να υπογραμμιστούν προς τα κράτη-μέλη και προσπαθώ να το κάνω συνέταξα την πρότασή μου ε, σε σχέση με ένα αριθμό εγγράφων μεταξύ των οποίων και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του προηγούμενου Νοεμβρίου και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που το ακολούθησε. Είχαμε επίσης μια προφορική ανακοίνωση του Συμβουλίου το Φεβρουάριο που δημοσιεύθηκε στις 17 Μαΐου και εγώ ε, δεν το έχω δει δημοσιευμένο βέβαια όπως καταλάβατε, εργάστηκα μόνο σε σχέση με αυτά τα οποία είχα ακούσει. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία ε, να μας προκαλέσουν το ενδιαφέρον. Είδα επίση και την έκθεση της ΕΦΣΑ για την θνησιμότητα των μέλισσών. Είναι μεγάλη έκθεση, αλλά αρκετά εύκολο να τη διαβάσει κανείς, αν και είναι εκατοντάδε σελίδες. Έχει σημασία να εξεταστεί η έκθεση αυτή για την θνησιμότητα των μελισσών, γιατί αυτά τα οποία θα συζητήσουμε ακόμα και σε οικονομικό επίπεδο εξαρτώνται από το πώς θα κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η επιστήμη αντιμετωπίζει τα θέματα. Και αν δεν γνωρίζουμε τον τρόπο αυτό, τότε είναι προφανές ότι θα υπάρξουν παρανοήσεις και στρεβλώσεις. Δεν σκοπό να σας διαβάσω τη γνωμοδότησή μου φυσικά, αλλά να πω ότι έχουμε εδώ να κάνουμε με πολλούς παράγοντες. Δεν υπάρχει ένα θέμα μόνο σχετικό με τις μέλισσες, το οποίο να οδηγεί στην μείωση του επίπεδου υγείας των μελισσών. Υπάρχουν πολλά θέματα και ο πληθωρισμός και η σόρευση όλων αυτών των προβλημάτων επιδρά την, τις μέλισσες με διαφορετικό τρόπο. Περιμένω τις αντιδράσεις των μελών γύρω από το θέμα. Λοιπόν, κλάες. Σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την συνάδελφο για τη σύντομη εισαγωγή στην έκθεσή της. Αληθεύει έχει λίγα στοιχεία που μπορεί κανείς να γράψει. Δεν μπορεί όλα να τα συντάξει και να τα γράψει όσα θα ήθελε. Όμως το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από πλευράς αρχής πολλά πράγματα θίγει και καλύπτει και νομίζω η πρόθεση που έχουμε ενώπιόν μας είναι η σωστή, η σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πραγματικά όλοι ότι οι μέλησες είναι το σημαντικότερο σε αυτό το στοιχείο. Χωρίς αυτές δεν θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε εμείς οι άνθρωποι. Ε, τα περισσότερα από τα δικά μας ενδυμικά φυτά εξαρτώνται από την γονιμοποίηση, από την ε, επικονίαση από τις, μύγες, από τις μέλισσες και όταν γνωρίζει κανείς ότι ε, τα μελίσια αυτά συνεισφέρουν και είναι πρόθυμοι πολύ να πληρώσουν κιόλας για την ύπαρξή τους ώστε να υπάρξει επικονίαση για να υπάρξουν τα φρούτα ε, είναι κάτι σημαντικό. Είχαμε και ένα ψήφισμα πριν από περίπου δύο χρόνια και ζητούσαμε αυστηρότερε προποθέσει για ένα πρόγραμμα δράση κατά τη θνησιμότητα των ε, μελισσών και την ε, ένταξη των ασθενειών των μελισσών στην ευρωπαϊκή κτηνιατρική πολιτική ω θέμα. Και χαιρετίζω την πρόθεση και πρωτοβουλία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα ίδια αναλυφθέντα μέτρα για την υποστήριξη των εθνικών μελισσοκομικών προγραμμάτων. Συχνά ωστόσο όμω επικεντρωνόμαστε εστιαζόμαστε στην σχέση μεταξύ πεδίο έντασης μεταξύ γεωργών και χρήσης φυτοκτόνων αφενός από πλευρά τους και των μελισσοκόμων από την άλλη και των συμφερόντων τους. Η πείρα έδειξε ότι ένα ευρύ φάσμα είναι το σωστό που πρέπει να ακολουθηθεί για την προστασία των μελισσών. Και εδώ ένα ευρύτερο φάσμα πρέπει να προσεγγίσουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε το θέμα της θνησιμότητας των μελισσών που είναι πολυσχηδές θέμα. Πρέπει πολλοί παράγοντες να δούμε ότι επηρεάζουν και πολλά θέματα επηρεάζουν την ε, ε, θνησιμότητα ή τη δυνατότητα επιβίωσης ε, των ζώων αυτών. Και πρέπει να δούμε σε σχέση με τις, τους διαφορετικούς παράγοντες όταν για παράδειγμα μόνο κράμβι ε, είναι το διαθέσιμο στις μέλισσες τότε δεν είναι καλό για την υγεία τους. Από την άλλη πλευρά συνεισφέρει και το κλίμα, η γενετική ε, προδιάθεση, ε, η καλλιέργεια, η προστασία των μελισσών από πλευράς επαγγελματιών μελισσοκόμων, η σωστή επαγγελματική προσέγγιση ε, και την απαγόρευση ή μη χρήση των απαγορευμένων ε, επικίνδυνων φυτοκτόνων. Γι' αυτό είναι σημαντικό από τη μία και άλλη πλευρά να προωθήσουμε τις γνώσεις και μεταξύ των ερευνητών, μεταξύ γεωργών και μελισσοκόμων να υπάρξει διευκόλυνση, κατανόησης και εξοικείωση με τα θέματα. Εκεί όπου λόγω εσφαλμένης χρήσης φυτοκτόνων υπάρχει θνησιμότητα μελισσών, η συνεργασία μεταξύ μελισσοκόμων και γεωργών πρέπει να ενταθεί και να προαχθεί ώστε να το αποφύγουμε αυτό. Χρειαζόμαστε όπως είπα, μια συνολική, ολιστική προσέγγιση και συντονισμένη προσέγγιση. Και σε αυτό ανήκει και η περαιτέρω στήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων μετά το 2013. Και εδώ, μια και υπήρξε η αναφορά μέχρι 2013, αυτές οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν. Καλύτερη πρόσβαση, πελασιμότητα στην ιατρική, στα φάρμακα, η προστασία των μελισσών είναι ακριβώς το κύριο, κυριότερο συμφέρον των ίδιων των γεωργών. Παλιότερα οι περισσότεροι γεωργοί εργαζόντουσαν, είχαν δραστηριότητα και ως μελισσοκόμοι. Και αν δούμε στη δική μας περιφέρεια, για παράδειγμα, 10-15 μελισσοκόμοι υπήρχαν εκεί. Σήμερα δεν υπάρχουν πια. Και υπήρχαν επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, πώς να το πω, που ως δευτερογενές τομέας, ε, δευτερογενής τομέας ε, ήταν πεδίο δραστηριότητας για τους ε, γεωργούς. Δεν έχουν εξοικειωθεί ή δεν έχουν πλέον ενδιαφέρον ή συμφέρον να ασχοληθούν με αυτά οι γεωργοί σήμερα. Πρέπει να μας προβληματίσουν όλα αυτά. Όλα αυτά είναι λόγοι για την μείωση των μελισσιών οι μέλισσες δεν είναι άγρια ζώα, δεν είναι άγρια πανίδα. Μπορεί να θεωρηθούν και κατοικίδια εντό εισαγωγικών, εξημερωμένα ζώα. Χρειάζονται προστασία και φροντίδα. Και είναι πολύ λίγοι εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται επαγγελματικά με τις μέλισσες. Οι νέοι μελισσοκόμοι και οι, οι ερασιτέχνες μελισσοκόμοι πρέπει πολύ περισσότερο να στηριχθούν και να προαχθούν. Αν θέλουμε να ασχολούνται με το επάγγελμα του μελισσοκόμου στο μέλλον και δεν θέλουμε να ε, πάψει πια αυτή η δραστηριότητα. Πρέπει να υπάρξουν κίνητρα για να ασχοληθεί κανεί με τι μέλισσε να γίνει μελισσοκόμο. Χρειαζόμαστε κατευθυντήριε γραμμέ στην Ευρώπη για τι βέλτιστε πρακτικέ και προγράμματα κατάρτιση των μελισσοκόμων. Είναι σημαντικό να τα τονίσουμε αυτά και η κυρία Γέρλινγκ το είπε και πριν από δύο χρόνια ήδη είχαμε και προτάσει για τα διαθετικά μέτρα για την προστασία των μελισσών στην αναθεώρηση της ε, οδηγίας για την προστασία των φυτών. Αυτά που εγκρίναμε εδώ στοχεύουν σε μια σωστή κατεύθυνση για την υπεύθυνη αντιμετώπιση των ε, μελισσών και τη σωστή χρήση των ε, φυτοφαρμάκων. Η νέα ε, ε, οδηγία για τις αδειοδοτήσεις θα αρχίσει να ισχύει και έτσι λοιπόν και για τα στοιχεία αδειοδότησης διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο. Και εδώ αναμένουμε μια βελτίωση των πραγμάτων που θα είναι προς όφελος και των μελισσών. Αναφέρεται ότι τα φυτοφάρμακα μόνο τότε μπορούν να, να χρησιμοποιούνται όταν δεν θα υπάρχει επικίνδυνη επίπτωση στις ε, μέλισσες ή δεν θα υπάρχουν οξύτερες επιπτώσεις στα μελίσια. Δηλαδή, συνάδελφοι, σε δύο εβδομάδες θα αρχίσει να ισχύει αυτή η οδηγία για τα φυτοφάρμακα και την προστασία σε σχέση με αυτά. Εδώ αναμένουμε να υπάρξουν και νέα κίνητα, νέες ε, ε, προσεγγίσεις. Αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη με αυστηρό πνεύμα να ελέγχουν και τις, ε, την αξιολόγηση κινδύνων να την πραγματοποιούν σε τακτά διαστήματα. Καμιά φορά οι φυστάμενες διατάξεις, κανονισμοί θα πρέπει όχι μόνο να λέμε ότι θα εφαρμόζονται και να ελέγχονται ως προς την εφαρμογή τους. Θέλω ολοκληρώνοντας να θέσω ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην ανακοίνωσή σας λέγεται ότι θα υπάρχει ένα εργαστήριο αναφοράς για τις ε, μέλισσες. Θα καταρτιστεί και θα διοριστεί και ήδη από το 2011 θα αρχίσει να ε, εργάζεται. Και πώς εργάζεται αυτό. Θα ήθελα να τα μάθω τα σχετικά. Ευχαριστώ. Thank you very much. Uh, next shadow is Děkuji, pane předsedo. Ehm, velmi stručně eh, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έκανε. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, σίγουρα, και χαιρετίζω και την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χωρίς ε, γενικές εισαγωγές θα ήθελα να αναφέρω συγκεκριμένα θέματα που θα ήθελα να συμπληρώσουμε. Κυρίως θα έπρεπε να αναφέρουμε, να τονίσουμε ότι μεταξύ των νέων ζυζανιοκτώνων, ε, ε παρασιτοκτώνων υπάρχουν πολύ δηλητηριώδεις ουσίες. Κάποιες από αυτές ε, θεωρούνται από τους πραγματογνώμονες ως λόγος εξόντωσης πάμπολων μελισσιών. Όσον αφορά αυτό θα ήθελα να αναφέρω και τον κίνδυνο που οι νεονικοτίνες αποτελούν. Αυτές οι ουσίες δημιουργούν προβλήματα στις μέλισσες και, στις, ε, και συνεχίζουν και παράγονται όμως στα κράτη-μέλη. Σε κάποια κράτη-μέλη έχουν όμως ωστόσο ήδη απαγορευτεί. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε συνολικά να απαγορευτούν πανευρωπαϊκά. Το άλλο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω είναι οι περιπτώσεις ακριβώς στις οποίες εκείνες το μέλι έχει ε, εκείνο ήδη μολυνθεί και οδηγεί στις ε, ε, περιπτώσεις απώλειας ολόκληρων μελισσιών. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η μόλυνση θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και θα πρέπει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής αυτή η επιμόλυνση. Αν ο ιός τώρα αυτός οδηγεί συνεισφέρει στην απώλεια των μελισσιών ή αν είναι ο κύριος λόγος και όχι μόνο ε, παρεμπιπτόντος συνεισφέρει στην ε, εξόντωσή τους πρέπει να διερευνηθεί και να ε, διαπιστωθεί άμεσα. Εν πάση περιπτώσει τα μέτρα πρέπει να ληφθούν να αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος χωρίς να αναμένουμε και να παραμένουμε αδρανείς. Πιστεύω ότι οι εισαγωγέ από την Κίνα πρέπει να ελέγχονται αυστηρότατα. Οι εισαγωγέ επίση και από άλλε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση στην ανάλυση των παραγόντων που αφορούν την ε, θνησιμότητα των μελισσών πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι πρόκειται για κοινωνικότατα έντομα. Οι μέλισσες είναι κοινωνικότατα έντομα. Δεν μπορεί ένας παράγοντας μόνο να θεωρηθεί ότι είναι υπεύθυνο για, ένα για ένα από αυτά τα έντομα, αλλά για το σύνολο του μελισσιού. Και γι' αυτό διαδραματίζουν αυτοί οι λόγοι ε, σημαντικό ρόλο για, το, για τα μελίσια που κινδυνεύουν. Πρέπει να συλλεγούν και περαιτέρω στοιχεία που θα δώσουν τη δυνατότητα να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα. Μέχρι τότε θα πρέπει η αρχή της πρόνοιας και πρόληψης ε, να ισχύει. Σας ευχαριστώ. Next speaker Grazie, Presidente. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνάδελφο Γκέρλινγκ για την εξαιρετική της ε, παρουσίαση, έθιξε κάποια θέματα στα οποία εμείς έχουμε αρμοδιότητες, η Επιτροπή αυτή έχει αρμοδιότητες για να εκφραστεί. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την σημαντική ανησυχία που υπάρχει για την αύξηση της ε, θνησιμότητας των μελισσών και των εντόμων που προχωρούν σε επικονιάσεις. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει σήμερα και όχι ότι μπορεί να υπάρξει στο οικοσύστημα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι υπάρχουν ήδη αρνητικές πλευρές αυτού του φαινομένου και όχι απλές κάποιες ανησυχίες. Επί της ουσίας, ένα μεγάλο τμήμα των προβλημάτων ε, είναι θα έλεγα ε, σαφές. Υπάρχουν παράσιτα τα οποία εξασθενούν το ανοσοποιητικό των μελισσών, η σπάνης κάποιων φαρμακευτικών παρεμβάσεων, οι κλιματολογικές αλλαγές που δημιουργούν αλλαγές στις συνθήκες των οικοτόπων και η εντατική γεωργία. Γι' αυτό λοιπόν υποστηρίζω και εγώ όπως ε, συγητή της Άλντε την πρόταση δημιουργίας ενός εργαστηρίου αναφοράς για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επιλογή ενός τέτοιου εργαστηρίου υπέρ της υγείας των μελισσών για να καταλάβουμε ποια είναι τα προβλήματα συγκεκριμένα και να τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά να κάνω μία παρέμβαση σε δύο σημεία τώρα κάπως πιο συγκεκριμένη. Η έκθεση λέγει ότι δεν υπάρχουν επιστημονικές αποδείξεις για το ότι οι γενετικά τροποποιημένοι μηχανισμοί όπως επίσης και ε, οργανισμοί, συγγνώμη, όπως επίσης και τα παρασιτοκτόνα επηρεάζουν αρνητικά τις μέλισσες. Θα ήθελα να πω ότι μπορεί να ελείπουν πράγματι ε, κάποιες επιστημονικές παρατηρήσεις και οι αλλαγές στις φυσικές ισορροπίες συμβαίνουν σε επίπεδο μακροπρόθεσμο και δεν μπορούν να εξεταστούν, να διαπιστωθούν, να ειδωθούν αυτό στιγμή. Συνεπώς λοιπόν οφείλουμε εμείς να προσπαθήσουμε να τροποποιήσουμε λίγο την έκθεση έτσι ώστε αυτή η λογική που προανέφερα, η προβληματική που ανέφερα να συμπεριληφθεί. Μιλάτε επίσης για έλλειψη επιστημονικών δεδομένων λόγω της χρήσης των σύγχρονων παρασιτοκτόνων. Θα πρέπει όμως να μην αγνοήσουμε ότι υπάρχουν ορισμένες καταστάσεις οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί και είναι γνωστές στην επιστημονική κοινότητα που διαψεύδουν αυτό το οποίο λέτε. Εδώ και δύο χρόνια κυκλοφόρησε το νέο ότι ένα μεγάλο, μια μεγάλη εταιρεία των, του Ηνωμένου Βασιλείου απαγόρευσε την πώληση 8 εντομοκτώνων παρασιτοκτώνων τα οποία πολλούσε λόγω της βλάβης που προκαλούν στις μέλισσες. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να σας προβληματίσουν, λέει στην εισηγήτρια ο κύριος Αουτζίας. Θα ήθελα να κλείσω Αναφερόμενο στις δεκόμενες χρηστές πρακτικές, στην έκθεση λέγεται ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ειδικό χαρακτήρας της, ε, ε, της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Θα πρέπει να καταλάβουμε εδώ σε τι αναφέρεστε. Η πλειοψηφία των παραγωγών ε, μελιού και ε, κύρου είναι μικρή παραγωγή και αντιπροσωπεύουν σαν μικρή παραγωγή το 90% του συνόλου των παραγωγών και 67% ε, του συνόλου των Ευρωπαίων παραγωγών σε επίπεδο μελισσοκομείας. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο θα πρέπει επίσης να μείνουμε. Θα ήθελα να αναφερθώ στον κανονισμό 1698 του 2005 για την υποστήριξη στην ανάπτυξη της υπαίθρου ο συγκεκριμένος αυτός κανονισμός ενθαρρύνει να βελτιστοποιηθούν οι συνθήκες για την γενική ευημερία του πληθυσμού και λέγει επίσης ότι δεν είναι δυνατόν να αναλυφθούν υποχρεώσεις οι οποίες να δημιουργούν προβλήματα ερεσιμότητας για τους καλλιεργητές, κτηνοτρόφους κτλ. Και το ίδιο συμβαίνει και με τους μελισσοκόμους δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συνθήκη η οποία να είναι ομοιογενοποιημένη για την ευημερία των μελισσών. Δηλαδή πως ένα σμάρι μελισσών ε, είναι σε καλή υγεία, ε, σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να κινητοποιήσουμε τις μορφές χρηματοδότησης οι οποίες είναι διαθέσιμες για άλλες γεωργικές δραστηριότητες. Νομίζω λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει ίσως να υπάρξουν κάποιες σκέψεις και αυτό νομίζω ότι ίσως είναι αρμοδιότητα συγκεκριμένη της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ, Keith Τέιλορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάθομαι στη θέση του Μισελ Ραβέιζη που είναι και σκιώδης ε, συγγήτρια ε, για αυτήν εδώ την έκθεση. Δεν μπορούσαν εδώ σήμερα δυστυχώς ε, τελευταία άρχισα να ασχολούμαι μαζί, με αυτό το ζήτημα. Θα ξεκινήσουμε με τις παρατηρήσεις που έχω προετοιμάσει και που έχω λάβει από τη Μισελ. Ο τίτλος «Μέλισσα» στην πρώτη σελίδα είναι μάλλον παραπλανητικός. Βεβαίως και οι μέλισσες αυτές παράγουν μέλι, όμως η αξία αυτή είναι οριακή σε σχέση με την αξία της ε, επικονίασης. Η συνολική ε, οικονομική αξία της επικονίασης ε, εκτιμάται στα 153 δις ευρώ. πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με, την, με, το, με τη συνολική οικονομική αξία της ε, αγροτικής παραγωγής το 2005. Ε, όμως, σε ό,τι αφορά την επικονίαση, η αξία ε, είναι περίπου 20 φορές η αξία όλων των ε, προϊόντων αυτών μαζί. Επομένως θα πρέπει να βάλουμε στην ε, πρώτη σελίδα ε, μέλη τη Παύλα Επικονιαστέ. Εδώ πέρα έχουμε μια πολύ σημαντική απειλή γιατί πολλές ε, καλλιέργειες ε, επικονιάζονται ε, από τις μέλισσες. 87 από τις 115 κύριες καλλιέργειες τροφίμων βασίζονται στην επικονίαση από μέλισσες. Και συγκεκριμένες πολύ σημαντικές καλλιέργειες όπως κακάο και καφέ συνέχιση των απολειών αυτών θα μπορούσε να έχει δραματικές επιπτώσεις ε, στο περιβάλλον μας, στην ε, αστική ανάπτυξη, ε, περιφερειακή ανάπτυξη μάλλον και την ε, επιστηστική ασφάλεια. Η ανακοίνωση της Επιτροπής παρουσιάζει μια καλή σύνοψη όλων αυτών των πτυχών που αφορούν την υγεία των μελισσών. Ωστόσο παραμένει μάλλον ασαφής και υπάρχουν ε, πολύ σημαντικοί κίνδυνοι εάν καταρρεύσει ο πληθυσμό των μελισσών και χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή ανακοίνωση. Θέλουμε σχέδιο δράση με στόχου. Και θα θέλαμε να ακούσουμε την απάντηση τη Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο γνωμοδότηση που μα παρουσίασε η Judy Gerling, ναι, συμφωνούμε πάνω κάτω με όσα είπε. Αλλά ειλικρινά, στην παράγραφο 5 δεν κατανοούμε ακριβώς ε, τον πραγματικό στόχο. Ε, παίζετε εδώ πέρα τον ε, δικηγόρο του διαβόλου ή το εννοείται σοβαρά. Στην παράγραφο 5 λέτε ότι δεν υπάρχουν ε, αδιάστατα στοιχεία ότι τα σύγχρονα παρασιτοκτόνα και γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί έχουν αρνητικές συνέπειες για τους πληθυσμούς μελισσών. Και μάλιστα μας λέτε ότι οι διαδικασίες ελέγχου είναι πολύ αυστηρές και στηρίζονται με, από μέτρα ε, ευαισθητικής ασφάλειας. Εμάς μας εκπλήσει αυτό που λέτε, γιατί σε όλα τα κόμματα υπήρξε συμφωνία σχετικά με την αύξηση της προστασίας των μελισσών από τα παριστοκτόνα στο πλαίσιο νέου κανονισμού για την έγκριση των παριστοκτόνων που υιοθετήθηκε το 2009. Στην παλαιότερη νομοθεσία που ακόμα ισχύει σήμερα, οι χρόνιες συνέπειες ε, στις ε, ε, ε, απικίες μελισσών δεν έχουν ακόμα διαρευνηθεί και οι συνέπειες των παραστοκτώνων σε αυτές. ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την, τις συνέπειες τους, σε ό,τι αφορά και το νέκταρ και τη γύρι τους. Το 2009 λοιπόν ε, καταφέραμε να ε, καλύψουμε αυτό το κενό. Θέσαμε ένα συγκεκριμένο κριτήριο βάση του κινδύνου που συμπεριλαμβάνει τις χρόνιες συνέπειες ε, και τις νύμφες μελισσών. Ζητήσαμε και από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει πρωτόκολλα μελέτης που λαμβάνει υπόψη και τη γύρι και τον έκταρ. Από όσο γνωρίζω εγώ, η Επιτροπή έχει δεσμευθεί ως προς αυτό και ε, δραστηριοποιείται ενεργά ε, για την αναθεώρηση αυτών των προϋποθέσεων. Όμως, σύμφωνα με τις ίδιες τις ε, προβλέψεις της, οι νέες προϋποθέσεις που θα, που θα υιοθετηθούν θα ισχύσουν μόλις το 2013-2014 όμως ε, σίγουρα δεν θα ισχύσουν αναδρομικά. Ε, θα αφορούν ε, αιτήματα για τις νέες δραστικές ουσίες. Με άλλα λόγια, ακόμα κι αν αυτές οι νέες προϋποθέσεις είναι απόλυτα επαρκείς, θα ισχύσουν θα μας πάρει ακόμα 10 χρόνια μετά το 2013-2014 μέχρι τα παραστοκτών αυτά να υποβληθούν σε μια αυστηρή διαδικασία έγκρισης στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Γκέρλινγκ. Και τα ε, μέτρα καθορισμού κινδύνου δεν είναι καθόλου επαρκή, γιατί στη Γερμανία, για παράδειγμα, ανακλήθηκε η αδειοδότηση αρκετών ε, ε, προϊόντων ε, σε περαιτέρω αξιολόγηση. Το να πούμε όμως ότι τα βαριστοκτόνα είναι ο μόνος παράγοντας που καταστρέφει την υγεία των μελισσών, ε, βεβαίως και δεν είναι ε, καθόλου σωστό. Αλλά το να αποκλείουμε και τα βαριστοκτόνα από τους παράγοντες κινδύνου που οδηγεί στην ε, εξάλληψη των μελισσών και να λέμε ότι όλα είναι υποέλεγχο, όπως λέει η κυρία Γκέρλινγκ στις παραγράφους 3 και 5, είναι κατά τη γνώμη μου εξίσου ανεύθυνο. Ε, έχουμε και την αρχή της πρόληψης που αναφέρθηκε. Τι συμβαίνει λοιπόν με αυτή την αρχή της ε, πρόληψης. από ό,τι φαίνεται την έχετε ξεχάσει. Έχουμε ένα αίτημα προς την κυρία Γκέρλινγκ να επανεξετάσει αυτή την γνωμοδότηση. Γιατί απέχει πολύ από την ε, ε, θέση όχι μόνο αυτής της Επιτροπής αλλά και του συνόλου του Κοινοβουλίου. Δεύτερον, ε, αντικειμενικά είναι λανθασμένη, εσφαλμένη βάση των συνεχιζόμενων αλλαγών στην σχετική νομοθεσία, οι οποίες όμως ε, θα γίνουν πολλά χρόνια μετά. Και τρίτον, είναι αντιπαραγωγικό να πούμε ότι η ασφάλεια δεν μπορεί να διαβεβαιωθεί ακόμα. Έτσι τρέχουμε τον κίνδυνο σωματικών αλλαγών, ε, μάλλον ε, της διακύβευσης σημαντικών αλλαγών κατά την αλλαγή της διαδικασίας αδειοδότησης των παραστοκτώνων. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Αγγέλη, και να σας ζητήσω να το επανεξετάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω το λόγο στον τελευταίο σκιώδη, την Καρτίκα Λιόταρντ, έχουμε μια περίεργη κατάσταση να αντιμετωπίσουμε. Μας τελείωσαν οι αντιπρόεδροι. Εγώ πρέπει να πάω στι διαπραγματεύσει ε, για την έκθεση, για την ετικετοθεσία που ξεκινάει στις 5. Σύμφωνα με τον κανονισμό, αν δεν υπάρχουν αντιπρόεδροι, Αυτό που πρέπει να αναλάβει την προεδρία είναι το παλαιότερο μέλος στην Επιτροπή. Και στην περίπτωσή μας είναι η Κρίστα Κλάες. Ε, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα ήθελα να δώσω την Προεδρία στην Κρίστα Κλάες. Καλή σας τύχη. Σε ευχαριστώ πολύ Καρλ Σλούιτα. Και μένα με πιάσε τώρα η μπάλα. Θα πηδήξω στο κρύο, στα κρύα βαθιά νερά να δούμε πώς θα μπορέσω να τα καταφέρω. Αλλά έχω και καλούς ε, από τη γραμματεία στο πλευρό μου. Λοιπόν, μπορώ να δώσω τον λόγο στην ε, σκιώδη συγγήτρια, συνάδελφό μας. Παρακαλώ, Ατίνκα. Σας ευχαριστώ, κυρία Κλάς. Και εγώ πρέπει σε αυτή τη συνεδρίαση, όπως και ο συνάδελφος Σλούτερ, να ε, μπορέσω να τα καταφέρω. Θέλω να, θέλω να πω το χαιρετίζω καταρχήν ότι συντάσσουμε μια έκθεση για τις μέλισσες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μέλισσες. Ήδη στο παρελθόν επανειλημμένα το Ευρωκοινοβούλιο είχε πει ότι ανησυχεί, ανησυχεί για τη θνησιμότητα των ε, των μελισσών και θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτό το πρώτο σχέδιο έκθεσης που μας ε, υπέβαλε και θα ήθελα ευχαρίστως να ανταποκριθώ στην πρόσκλησή της να προσπαθήσουμε αναμεταξύ μας το κείμενο αυτό να το βελτιώσουμε όσο γίνεται περισσότερο γιατί υπάρχουν μια σειρά, ε, μια, ε, αρκετές πτυχές ε, που πρέπει να καλυφθούν. Θα ήθελα καταρχήν πάλι να παρακαλέσω την εισηγήτρια να ξαναδεί τον τίτλο αναφέρεται λέει για την υγεία των μελισσοπαραγωγών μελισσών. Αυτό θα μπορούσε να αναφέρει ότι καμιά φορά έχουν κάποιο ακριολόγημα ή μικροαρρωσταίνουν, ψηλοαρρωσταίνουν οι μέλισσες, αλλά αυτό περί το οποίο πρόκειται ουσιαστικά είναι <clears throat> μαζική θνησιμότητα των ε, μελισσών. Περί αυτού πρόκειται και όταν συντάσσουμε μια έκθεση στην οποία εκφράζουμε τις ανησυχίες μας ως Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να αντανακλάτε και στον τίτλο της έκθεσης αυτό. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω λοιπόν να ληφθεί υπόψη. Θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες ώστε να τροποποιηθεί ο τίτλος και να προσαρμοστεί θνησιμότητα των μελισσών και αντιμετώπιση της, ώστε με σαφήνεια να περιγράφεται το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Όποιος, όπως αναφέρθηκε από την ίδια, τα αίτια της νησιμότητας αυτής είναι ένας συνδυασμός αρκετών αιτίων και παραγόντων. Το αναφέρει και υπό αντίστοιχο εδάφιο αναφέρεται αυτό διεξοδικότερα ότι υπάρχει ένας μήκητας, υπάρχει ένας ιός, σίγουρα. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε ακριβώς γιατί έχει τέτοιες μαζικές διαστάσεις αυτή η θνησιμότητα των μελισσών και νομίζω δεν επαρκεί. Δεν επαρκεί όταν λέμε ότι τα φυτοκτόνα ε, και ε, τα διάφορα παρασιτοκτόνα και τα λοιπά ότι πρέπει με κάθε προσοχή να χρησιμοποιούνται γιατί είναι επικίνδυνες ουσίες. Εντάξει, ούτως ή άλλως. Αυτό αφορά και την ασφάλεια τροφίμων και την εξέτασή τους ως προς την ασφάλεια τροφίμων. Πρέπει να πούμε όμως σαφέστατα στην έκθεσή μας ότι θέλουμε να γίνουν έρευνες ε, για τις επιπτώσεις που έχουν στη θνησιμότητα των μελισσών επιπτώσεις ε, των φυτοκτόνων και ζυζανιοκτόνων και παρασιτοκτόνων στη θνησιμότητα των ε, μελισσών. Αλλά επίσης ε, και ακτινοβολία των κεραιών όσον αφορά τις μέλισσες, γιατί πολλές φορές αυτή η ακτινοβολία παρακολύει τις μέλισσες, δεν μπορούν να βρουν το δρόμο τους να επιστρέψουν στις κυψέλες τους, στα μελίσια. Και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και όχι μόνο εμπορικά πρέπει να δράσουμε για να προστατευτούν οι μέλισσες, αλλά έχουμε Θα πρέπει λοιπόν ο εισηγητή ακόμα να εργαστεί περισσότερο, η μάλλον να εργαστεί περισσότερο σε αυτό και ελπίζω να έτσι να μπορέσουμε να καταστήσουμε ακόμα πιο ισχυρή αυτή τη νομοδότηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο γύρος των σκιωδών εισηγητών ολοκληρώνεται. Παρακαλώ τώρα εσείς θα λάβετε τον λόγο. Thank you very much, sir. Uh, I would like... Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την έκθεσή της. Θα ήθελα να υπογραμμίσω τρία θέματα τα οποία έκαναν άλλωστε και οι συνάδελφοι. Το θέμα τι γίνεται με τα νεονικοτινοειδή αυτή τη νέα μορφή εντομοκτώνων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, τίθε είναι σε κάτι που απασχολεί πολύ κόσμο και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από πάρα πολλές χώρες. Γιατί μερικές φορές έχουν θανατηφόρες συνέπειες αυτά τα εντομοκτώνα. But other like bird Γνωρίζουμε ότι η Γερμανία, η Σλοβενία και η Γαλλία έχουν ήδη απαγορεύσει τέτοιου είδους εντομοκτώνα και είναι καιρός πλέον και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση. Ταυτόχρονα έχουμε το θέμα των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. The BT, ε, the, the... Ιδιαίτερα στα BT. Οι ουσίες αυτές έχει αποδειχθεί μετά από μια μελέτη Γάλλων και Μεξικανών επιστημόνων ότι επηρεάζουν τη μνήμη και το ανοσοποιητικό των μελισσών. Οι ουσίες BT στα αγγλικά. Δεν έχουμε πολλές μελέτες. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί σε σχέση με την επιρροή των ουσιών αυτών στις, στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία με τα οποία κινούνται οι μέλισσες. Ε, υπάρχουν περιορισμένες μελέτες, είναι αλήθεια, αλλά αυτό δεν είναι λόγος να μείνουμε αδρανείς. Θα πρέπει να πάρουμε μια κάποια απόφαση. Ή γιατί έχουμε την υποχρέωση να το κάνουμε σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, με την αρχή της πρόληψης, και ώσπου να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα τότε θα πρέπει να λάβουμε περιοριστικά μέτρα, όχι μόνο για να υπερασπίσουμε το μέλι και τις μέλισσες, αλλά τη γεωργία γενικότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ κυρία Σένη. Επόμενη και τελευταία, η κυρία Λιζαμπέτα Λουκασέφσκα παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ η ίδια να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, να ευχαριστήσω για το γεγονός ότι συνέταξε αυτή τη σημαντική έκθεση και αποσαφηνίζει, θέτει στο σωστό πλαίσιο τα σημαντικά αυτά θέματα. Η θνησιμότητα το ποσοστό θνησιμότητα των μελισσών είναι σοβαρότατο πρόβλημα. Θέτω το ερώτημα, αυτό το πρόβλημα δεν τίθεται ε, αρκετά όψιμα, δεν έχουμε καθυστερήσει. Σε σχέση με το σημείο 3 και άλλα, ε, ε, όταν αναφέρονται τρία, τρεις συντελεστές, τρεις παράγοντες που συνεισφέρουν για, στη θνησιμότητα αυτή των μελισσών, ε, με τους μελισσοκόμους όταν έχετε κανεί σε επαφή και όταν ε, εξοικειώνεται με αυτά τα θέματα, κάποιοι από τους προλαλήσαντες ανέφεραν ότι πρόκειται για ερασιτέχνες, ότι είναι ερασιτέχνες μελισσοκόμοι που δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις Πιστέψτε μου, μετα, μεταφέρονται οι γνώσεις από τη μία γενεά στην άλλη. Και αν αναφέρονται αυτοί οι τρεις παράγοντες, αυτοί που προαναφέρθηκαν, δεν θα υπήρχε, αν ελαμβανόντουσαν υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία, δεν θα υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Λένε οι μελισσοκόμοι, το πρόβλημα έγκυται μεταξύ άλλων, κυρίως στο εξή ζήτημα, στο ότι τα αίτια βρίσκονται, οφείλονται στο ότι φυτοκτόνα και παρασυτοκτόνα χρησιμοποιούνται. Γι' αυτό έχω ιδιαίτερες επιφυλάξεις όταν υπό το εδάφιο 5 βλέπω ότι δεν υπάρχουν λέει τεκμήρια και δεν υπάρχουν αποδείξεις για το ότι οι φυτοκτόνα και παρασυτοκτόνα έχουν άμεση επίπτωση στη θνησιμότητα των μελισσών. Δεν μπορεί να είναι έτσι, διότι πιστεύω τους μελισσοκόμους που εμπειρικά παρακολουθούν αυτή, αυτή, την ε, μάστιγα τις ε, μέλισσες να εξοντώνονται και υπάρχει σχέση αιτίου και αιτιατού. Τα φυτοκτόνα και τα παρασιτοκτόνα είναι αίτια λοιπόν. Πολλοί τόνισαν ότι οι μελισσοπαραγωγές μέλισσες έχουν, μελισσοπαραγωγοί μέλισσες έχουν μεγάλη σημασία για μας, την κοινωνία μας και το περιβάλλον. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το ότι οι επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με τα θέματα αυτά είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά, όχι μόνο στα αίτια, γιατί δηλαδή με άλλα λόγια οι μέλισσοπαραγωγές, μέλισσες ε, αθνείς που πεθαίνουν, αλλά να δούμε και τη διαδικασία της αδειοδότησης των φυτοκτόνων και των παρασιτοκτόνων. Όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν και να εξεταστούν σε βάθος, διότι άσχετα από το, τις γνώσεις των μελισσοκόμων, όλα αυτά αλλοιώνονται, αλλάζουν σήμερα. Ακόμα και τα παραστοκτόνα και τα φυτοκτόνα. Χρειάζονται περισσότερες γνώσεις ε, οι μελισσοκόμοι. Χρειάζονται κατάρτιση. Χρειάζονται και οικονομική υποστήριξη για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων ώστε να μπορέσουν να βασίζονται, να μπορούν να βασίζονται στην υποστήριξη. Να βασίζονται σε μια υποστήριξη και να μην είναι τα ε, παραπέδια, α το πω έτσι, σε σχέση με τους γεωργούς όσον αφορά τη στήριξη. Σας ευχαριστώ, Λουκασένκα. Θα δώσω τον λόγο στην Επιτροπή, για την Επιτροπή ο κύριος Λαντομάντα παρίσταται. Θα ήθελα να τον παρακαλέσω να τοποθετηθεί σε σχέση με τις αμφίσιμες, αμφίροπες αυτές ε, τοποθετήσεις των συναδέφων για τα πανστιοκτώνα και ζυζανιοκτώνα και να δούμε σε σχέση με τον νέο κανονισμό, με τη νέα οδηγία που θα αρχίσει να ισχύει, αν έχουμε κάποια πράγματα ρυθμίσει ή πρέπει να ξαναρυθμιστούν, να ρυθμιστούν και να προσαρμοστούν. Ευχαριστώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω τις δράσεις τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει και αυτές που σκοπεύει να αναλάβει στο προσεχές μέλλον σχετικά με την υγεία των μελισσών. Καταρχάς έχουμε ορίσει ένα νέο εργαστήριο αναφοράς για την υγεία των μελισσών. Έγινε με τον τακτό τρόπο, όπως προβλέπει η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πρόκειται για το εργαστήριο «Ανσες» στη Σοφία Αντίπολη της Νότιας Γαλλίας από την 1η Απριλίου του 2011 και έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση κατά 250.000 ευρώ για τους πρώτους τρεις μήνες δραστηριότητας. Έχουμε ξεκινήσει ορισμένες δραστηριότητες σχετικά με την κατάρτιση των επισήμων των κρατών μελών, των υπαλλήλων των κρατών μελών και των ιδίων των μελισσοπαραγωγών. Έχουμε ξεκινήσει επίσης και προγράμματα αναφοράς υποστήριξης των εθνικών προγραμμάτων ε, μελισσοκομείας. Το θέμα είναι ποιες είναι οι αιτίες της θνησιμότητας των μελισσών. Δεν είναι εύκολο να το πούμε αυτό. Αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε με την υποστήριξη ακριβώς του εργαστηρίου αναφοράς είναι να ξεκινήσουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα ελέγχου το οποίο θα γίνει αντικείμενο διαχείρισης από τα κράτη-μέλη για να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Θα πρέπει να ενισχυθούν φυσικά τα κριτήρια για την έγκριση ε, κάποιων εντομοκτώνων. Αυτό είναι τμήμα του νέου νομοθετικού πακέτου σχετικό με τα εντομοκτώνα συνολικότερα. Εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε με σωστό τρόπο τη νέα νομοθεσία η οποία θα τεθεί σε ισχύ σε σταδιακή φάση. Μιας και πρόκειται για ένα συγκεκριμένο θέμα, η συνάδελφος Φραντσέσκα Ρένα θα μπορούσε ίσως να προσθέσει κάποια επιπλέον τεχνικά στοιχεία. Θα ήθελα να υπογραμμίσω επίσης ότι είναι εν διαδικασία η αναθεώρηση των ιατρικών και φυτοφαρμάκων ε, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την υγεία των μελισσών. Αυτό είναι βασικό και για την υγεία των μελισσών, αλλά και για τη διασφάλιση του ότι το μέλι το οποίο παράγεται να περιλαμβάνει επαρκή ε, ή μάλλον όχι υπερβολικές ποσότητες και ποσοστά φαρμάκων και φυτοφαρμάκων. Η Επιτροπή επανεξετάζει το σύνολο της νομοθεσίας των φυτοφαρμάκων, μεταξύ των οποίων και αυτών που προορίζονται για τις μέλισσες. Λοιπόν, αν δεν σας πειράζει η Πρόεδρε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στη συνάδελφο Σέτα για να προσθέσει κάτι για τα εντομοκτώνα. Ευχαριστούμε πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο συνάδελφος Αρσένης έχει μια σύντομη επερώτηση. Σύντομα όμως παρακαλώ. I uh, Ήθελα να ακούσω αρχικά τη δεύτερη παρέμβαση της Επιτροπής. Το ερώτημα όμως είναι αν υπάρχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία ολοκλήρωσης της ε, ε έρευνας, αν έχουμε δεδομένα ή τουλάχιστον έχουμε δεδομένα για το τι προκαλεί τον θάνατο των μελισσών, αλλά αιδάλλως πού μπορούμε να εφαρμόσουμε την αρχή της πρόληψης. Ναι, στην απάντηση παρακαλώ να ενταχθεί και αυτό το θέμα. Παρακαλώ έχει τον λόγο η Επιτροπή. Το πιλωτικό σχέδιο το οποίο θέλει να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα κράτη-μέλη για τον έλεγχο ε, που θα πρέπει να γίνει θα διαρκέσει τρία χρόνια. Αυτό δεν είναι κάτι βέβαια το οποίο συνδέεται αποκλειστικά με τον εντοπισμό του προβλήματος ή των προβλημάτων που έχουν σχέση με τα εντομοκτώνα. Με άλλα λόγια, δεν είναι σαφές ότι μέσα σε τρία χρόνια θα είμαστε σε θέση εμείς να αξιολογήσουμε αποτελεσματικά κατά πόσον ε, τα εντομοκτώνα, τα παρασιτοκτώνα επηρεάζουν ε, το σύνολο του πληθυσμού των μελισσών. Δεν είναι δυνατόν να σας δώσω ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για αυτού του είδους ε, την ερώτηση. Αλλά σχετικά τώρα με την χρήση της αρχής της πρόληψης σε σχέση με τα παρασιτοκτόνα, η συνάδελφος είναι έτοιμη να πάρει το λόγο. Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι πράγματι ότι διαμορφώνουμε νέες απαιτήσεις για τα δεδομένα για τα παρασιτοκτόνα για να αυστηροποιήσουμε τα κριτήρια έγκρισης και των ουσιών και την αδειοδότηση κυκλοφορίας των συγκεκριμένων προσκευασμάτων. Αυτές οι απαιτήσει για πρώτη φορά περιλαμβάνουν και απαιτήσει για την αξιολόγηση του λεγόμενου χρόνιου κινδύνου χρήσης ε, των ε, παρασιτοκτόνων. Αυτό δεν περιλαμβάνεται στην υπάρχουσα νομοθεσία. Ζητάμε λοιπόν στοιχεία και για την καταμέτρηση ε, των επιπτώσεων σε δευτερευόντων ε, επιπτώσεων, όχι μόνο ε, στις μέλησες αλλά γενικότερα. Αυτές οι απαιτήσει, αυτά τα νέα δεδομένα θα απαιτηθούν από το τέλος του 2013 και ελπίζουμε να εφαρμοστούν άμεσα από το τέλος του 2013 όχι μέσα σε μια σταδιακή εφαρμογή δεκαετίας, αλλά άμεσα θα πρέπει να εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη όταν εκδίδονται ε, νέες αδείες για προϊόντα φυτοπροστασίας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υιοθετηθεί μια ουσία ε, η οποία αδειοδοτείται για μία δεκαετία. Επί της αρχής δεν πρόκειται να επαναξεταστεί η εγκυρότητα αυτής της άδεια εφόσον δεν υπάρχουν νέα δεδομένα. Αλλά από εδώ και πέρα η αδειοδότηση νέων προϊόντων θα γίνεται επί τη βάση των νέων απαιτήσεων ε, χορήγησης στοιχείων για τα νεονικοτινοειδή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανεξετάσει τα κριτήρια έγκρισης τις απαιτήσει έγκρισης το 2010. Είχαμε μια οδηγία, την 21 του 2010, και ζητάμε στην οδηγία αυτή από τα κράτη-μέλη να κάνουν συγκεκριμένα προγράμματα ελέγχου για νέο νοικοτινοειδή, για την οξιολόγηση των εντομοκτώνων στη δημόσια υγεία. Ελπίζουμε να έχουμε τα πρώτα στοιχεία μέχρι το τέλος του 2011 αν και δεν ξέρουμε ακριβώς αν θα μπορέσουμε να πάρουμε αποφάσεις με βάση τα συγκεκριμένα αυτά δεδομένα. Αλλά βασιζόμενοι στην αξιολόγηση των πληροφοριών τις οποίες θα λάβουμε από τα κράτη-μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει τις συνθήκες έγκρισης προϊόντων αυτού του τύπου νεκοτινοειδών. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να εφαρμόζουμε την αρχή της πρόληψης όπως και το κάναμε άλλωστε μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε πολύ για τις πρόσθετες αυτές επεξηγήσεις. Η κυρία εισηγήτρια θα λάβει για να ολοκληρώσει τον λόγο και πάλι παρακαλώ. Thank you. Um... Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα γενικά για να μην αναφερθώ σε όλα τα σχόλια σε μία προσημείο. Αρχικά να υπενθυμίσω στην Επιτροπή ε, το καθεστώς αυτής της γνωμοδότησης. Πρόκειται για μία γνωμοδότηση για, ε, βάση ε, ιδίας πρωτοβουλίας ε, της Άγκρη. Τα ζητήματα αυτά στα οποία αναφέρομαι λοιπόν ε, αφορούν κυρίως ε, την Επιτροπή Γεωργικών Υποθέσεων. Και μάλλον θα γνωρίζετε ότι εγώ συζητούσα για αρκετό καιρό μαζί με τον πρόεδρο εκείνης της Επιτροπής για να αναλάβουμε από κοινού την ευθύνη, αλλά δεν συμφωνήθηκε αυτό. Ε, ό,τι θέση για να πάρουμε για την νομοδότηση θα πρέπει να τη λάβουμε έχοντας αυτό κατά νου. Επομένως το θέμα δεν είναι να αλλάξουμε τον τίτλο ή κάτι τέτοιο. Ε, μάλλον ε, δεν είναι, ε, μάλλον άσχετο αν θέλετε είναι αυτό εδώ. Το θέμα είναι ότι εδώ οι μέλισσες ε, αναφέρονται εδώ σε αντιδιαστολή με τους άγριους ε, επικονιαστές. Ανέφερα βέβαια σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τους άγριους επικονιαστές. Αλλά δεν πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό, σε αυτή την επιτροπή, γιατί δεν είναι εδώ αυτό το πεδίο εφαρμογή της, ε, νομοδότηση. νομοδότησης. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο ξεκάθαρο σημείο είναι το σημείο των ε, νέων νοικοτενοειδών. Ε, πολλά ακούστηκαν για αυτό το ζήτημα και από τον Κίθ και από άλλους για την αποδεδειγμένη θανατηφόρα τους δράση. Με πολύ προσοχή συνέταξα το σημείο 5 της ε, γνωμοδότησής μου και αυτό γιατί η διατύπωση αυτή ε, συνάδει απόλυτα με αυτό που μας έχει παρουσιαστεί και, στις, ε, και στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και υιοθετήθηκε ε, στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου τον προηγούμενο Νοέμβριο. Ξέρω ότι έχουν γίνει ε, παρουσιάσεις από ανθρώπους που έχουν κάνει μικρές μελέτες και υπάρχουν ενδείξεις ότι ίσως ε, υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι ουσίες αυτές επηρεάζουν. Δεν λέω το αντίθετο. Εντάξει, σίγουρα είναι τολμηρή η διατύπωση, αλλά μπορείτε να αποβάλλετε τροπολογίε. Αυτό που θέλω να σα ε, παρακαλέσω όμω να μην αντιδράσετε μόνο σε αυτό. Γιατί η γνωμοδότηση αυτή αποτελεί μια ευκαιρία να επηρεάσουμε την Επιτροπή Γεωργικών Υποθέσεων. Στι ε, συνεδριάσει μα, κυρίω για την κοινή γεωργική πολιτική, πάντα λέμε πώ μα ανησυχεί το γεγονό ότι δεν υπάρχει ε, διασφαλισμένη χρηματοδότηση για τον τομέα μετά το 2013. Αυτό προκύπτει κυρίως από την ε, ε, κοινή γεωργική πολιτική. Και έτσι μπορεί να χάσουμε μια πολύ σημαντική ευκαιρία. Ορισμένα ζητήματα που αφορούν τη βιοπικιλότητα, για παράδειγμα, ε, είναι πολύ σημαντικό να μεταφέρουμε την άποψή μας στα ζητήματα αυτά στην Επιτροπή Γεωργικών Υποθέσεων. Και όλο αυτό το ζήτημα, για να επανέλθω στους ε, γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς, ίσως να αφορά και τις μονοκαλλιέργειες αυτό. Γιατί καλλιεργούνται, εμφανίζονται κυρίως μονο, ε, μονοκαλλιέργειες και οι μέλισσες, στις μέλισσες δεν αρέσουν οι μονοκαλλιέργειες, τους αρέσει η ποικιλία. Υπάρχουν λοιπόν πολλά διαφορετικά ζητήματα. Λαμβάνω υπόψη βέβαια όσα αναφέρθηκαν εδώ, αλλά παρακαλώ να υπάρχουν σχόλια βάσει ε, επιστημονικών ενδείξεων και όχι ε, συναισθηματικές αντιδράσεις μην εστιάζετε μόνο σε αυτό, εξετάστε και το υπόλοιπο της νομοδότησης, γιατί εδώ πέρα έχουμε μια ευκαιρία να μιλήσουμε κατευθείαν στους συναδέλφους μας στην ε, ε, Επιτροπή Άγκρη και να τους ε, εκφράσουμε τις απόψεις μας για αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα στο πλαίσιο της, του γεωργικού τομέα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκάρλινγκ. Η συζήτηση έτσι ολοκληρώθηκε για απόψε. Υπάρχει ευκαιρία κατάθεση τροπολογιών από όλους. Προθεσμία κατάθεση είναι η 15η Ιουνίου. Έχει λίγο πάει πιο πίσω, διότι η Επιτροπή Γεωργίας ως η αρμόδια Επιτροπή θα πρέπει να ψηφίσει πιο πριν. Μετά 13 Ιουλίου και αναμένουμε τις τροπολογίες 13 Ιουλίου η Ολομέλεια. Περνάμε στο σημείο 20 της ημερήσιας διάταξης. Είναι αυτό η έμεση αλλαγή χρήσης γης υποσυζήτηση ως θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ανακοίνωσή της του Δεκεμβρίου 2010 θα επεξηγήσει σχετικά και δίνω τον λόγο στην αρχή πρώτα-πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι παρόν, έχει τον λόγο λοιπόν, παρακαλώ. Thank you very much, Madam Chairman. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν είμαι ο Φιλιππών, είμαι ο Φρανς Χαρστίν. Ο Φίλιππον είναι ακριβώς δίπλα μου. Αυτός, ε, αυτό το φάκελο τον χειρίζονται δύο γενικές διευθύνσεις ε, της Επιτροπής, Γενική Διεύθυνση Ενέργεια και Κλιματικής ε, δράση. Εκπροσωπούμε αυτές τις δύο γενικές διευθύνσεις λοιπόν. Θα σας παρουσιάσουμε από κοινού τα, τα σχολιά μας σήμερα. Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε αυτή τη δυνατότητα. Είναι η δεύτερη φορά νομίζω που εξετάζουμε αυτό το θέμα ε, στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή αυτή μάλλον. Είχαμε μια ανταλλαγή απόψεων ε, πέρσι τον Νοέμβριο. Και από τότε, όπως είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε, η ε, Επιτροπή έχει παρουσιάσει την έκθεσή της στις 22 Δεκεμβρίου. Και με τα χαράς να σας την παρουσιάσουμε εδώ σήμερα. Ενημερωτικά να σας εξηγήσω περί τίνος πρόκειται είναι ένα θέμα το οποίο ανέκυψε εξαιτίας του πακέτου «Ενέργεια και κλίματος που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Περιλαμβάνει έναν αριθμό ε, στόχων. Πρώτον, το στόχο του 20% για το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το 2020. 10% το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, στις μεταφορές, μέχρι τότε και πάλι την ίδια προθεσμία. Επιπλέον, στην ποιότητα καυσίμων, στην οδηγία ποιότητα καυσίμων, στόχος για τη μείωση των εκπομπών ή μάλλον ε, αερίων του θερμοκηπίου κατά 6% μέχρι το 2020. Με αυτού του στόχου λοιπόν έχουμε ισχυρά κίνητρα για την απομάκρυνση από την κατανάλωση άνθρακα ε, σε αρκετούς τομείς, μεταξύ των οποίων και, το, και τις μεταφορές. Και σε αυτό θα συμβάλλουν ιδιαίτερα τα καύσιμα κατά τη γνώμη μας και αυτό έχει υπεβεβαιωθεί ε, από τα σχέδια που έχουν υποβάλει τα κρατημέλη υπό την ε, οδηγία για την με πηγές ενέργειας. Και εκεί μας έχουν εξηγήσει πώ ακριβώς θα ε, στόχο για παράδειγμα το 10% στι μεταφορέ. Πολύ σημαντικό τμήμα ε, των στόχων αυτών θα επιτευχθεί μέσω της χρήσης των βιοκαυσίμων. Αυτές οι δύο οδηγίες λοιπόν περιλαμβάνουν πολύ αυστηρά κριτήρια βιωσιμότητας για, τον, ε, για τους τύπους βιοκαυσίμων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη αυτών των στόχων. Τα κριτήρια αυτά αφορούν ε, ε, στις επιδόσεις αυτών των βιοκαυσίμων σε ό,τι αφορά τα αέρα του θερμοκηπίου, ποια φυτά μπορούν να μετα, μεταποιηθούν, μετατροποποιηθούν για να χρησιμοποιηθούν ως ε, βιοκαύσιμα. Και από πλευράς βιοπικιλότητας βέβαια. Ε, δηλαδή υπάρχουν εκτάσεις, ε, εδαφικές εκτάσεις που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αυτό το σκοπό. Ωστόσο, κατέστη ξεκάθαρο ότι υπάρχει θέμα με την έμεση αλλαγή της χρήσης της γης και γι' αυτό ε, ε, κληθήκαμε να υποβάλουμε έκθεση για αυτό το ζήτημα μέχρι τα τέλη του προηγούμενου έτους, πράγμα που πράξαμε. Για να κατανοήσουμε αυτό το θέμα, αυτό γιατί είναι, είναι ένα αρκετά περίπλοκο θέμα και ίσως είναι καλό να διευκρινίσουμε τι τίνος πρόκειται. Στην πράξη, αν έχουμε μία κατάσταση όπου έχουμε ε, απόθεμα ζωοτροφών ε, βιοκαυσίμων που ε, τροποποιείται από ένα άλλο καθεστώς, από άλλη χρήση, αυτό θεωρείται ότι πληρεί τα κριτήρια. Ωστόσο, άμα καλλιεργείται σε σε υπάρχουσε καλλιέργειες μπορεί έτσι να, υποκαταστήσει άλλε καλλιέργειε. κάτι που μπορεί να οδηγήσει στην ε, μετατροπή ε, γη ε, σε αγροτικέ καλλιέργειες. Αυτό εμεί χαρακτηρίζουμε ω έμεση αλλαγή χρήση γης. Αν αυτό συμβεί, αυτό θα φανεί μέσω αλλαγής της ζήτηση για αγροτικά αγαθά και τα αποκατάστατά τους στην παγκόσμια αγορά. Πώ μπορούμε να γνωρίζουμε αν συμβαίνει πράγματι κάτι τέτοιο. Πρώτα απ' όλα το είπαμε ξεκάθαρα στην έκθεση του Δεκεμβρίου. Συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αυτού του φαινομένου είναι ότι δεν μπορεί να παρατηρηθεί αμέσως ή να μετρηθεί αμέσως και έτσι ο μόνος τρόπος να το παρατηρήσουμε είναι μέσω τη χρήσης οικονομικών προτύπων. Και η Επιτροπή πράγματι έχει αναλάβει τέτοια εγχειρήματα τα οποία αναφέρουμε και στην έκθεση του Δεκεμβρίου. Πολύ λεπτομερώς. Επιπλέον έχουμε θέσει αυτές τις ε, εκθέσεις στη διάθεση ε, οποιοδήποτε ενδιαφέρεται. Το συμπέρασμα ήταν ότι η έμεση αλλαγή χρήσης γης υπάρχει, υφίστατος φαινόμενο, ταυτόχρονα όμως υποδεικνύουμε αρκετές ε, ελλείψεις και αβεβαιότητες ε, που σχετίζονται με αυτά τα πρότυπα. Ε, αναλύσαμε και τις διεθνείς εξελίξεις. Εδώ όμως θα δώσω το λόγο στον ε, συνάδελφο Φίλιπ για να συνεχίσει. Ευχαριστώ, Χάντς. Όπως εξήγησε ο Χάνς, ε, το θέμα αυτό χειριζόμαστε από κοινού. Οι δύο γενικέ διευθύνσει είναι περίπλοκο το ζήτημα και βεβαίω ο βαθμό συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών μα ε, είναι αρκετά υψηλό. Ούτω ώστε να σημειώνεται πρόοδο σε αυτό το φάκελο. Ε, η έκθεση αυτή εστίασε ιδιαίτερα στι διεθνεί πτυχέ ένα νέο πεδίο εργασιών αρκετές, ε, αρκετά κρατημέλη αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα της έμεσης αλλαγής χρήσης γης και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην ε, έκθεση. Πρώτα είδαμε την εμπειρία των ΗΠΑ τόσο σε ομοσπονδιακό και σε, και σε... Ε, τόσο σε ομοσπονδιακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πολιτιών γιατί σε ομοσπονδιακό επίπεδο προσπάθησαν να καθορίσουν ε, τον αντίκτυπο της έμεσης αλλαγής, αλλά και σε επίπεδο πολιτιών, στην Καλιφόρνια. Εκεί και πάλι συμπεριλαμβάνεται στην νομοθεσία τους. Σε αυτό το τμήμα ε, ε, εξετάσαμε και άλλα μέτρα, και άλλες μορφές μέτρων εξετάσαμε τι συμβαίνει στη Βραζιλία, όπου δημιουργούνται αγροοικονομικές ζώνες, αλλά και στην Αργεντινή, ε, όπου σταματάει η λοτομία μέχρι να ληφθούν νέα μέτρα. Τώρα, για, σε επίπεδο συντονισμού, και πάλι κοιτάξαμε σε, ε, τι συμβαίνει σε επίπεδο εταιρικών σχέσεων σε αυτόν τον τομέα. Αρκετά κράτη-μέλη συμμετέχουν, ε, μεταξύ των οποίων και η Βραζιλία και η Αργεντινή. Και βλέπουμε τι μπορεί να γίνει εκεί σε επίπεδο συντονισμού σε διεθνές, στο διεθνή χώρο. Συνοψίσαμε και τι πληροφορίες που λάβουμε από ενδιαφερόμενα μέρη. Υπήρξαν, ε, υπήρξε μια σειρά διαβουλεύσεων με τα ενδιαφέρομενα μέρη καθ' όλη αυτή τη διαδικασία, το 2009 αρχικά και μετά το 2010. Και εδώ συνοψίζουμε τα κύρια ε, συμπεράσματα. Για παράδειγμα, ε, από το εγχείρημα του 2009 έπαιξαν 71 απαντήσεις, στη διαβούλευση του 2010 145 απαντήσεις. Ε, το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο στην Ίσπρα Συγκάλεσε μια συνεδρίαση ε, εκεί ε, ε, για ανταλλαγή απόψεων και, και αυτό αναφέρεται εδώ, συνοψίζεται και υπάρχει και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής. Αντλήσαμε και ορισμένα συμπεράσματα από όλο αυτό το εγχείρημα, όπως ανέφερε και ο Χάνς. Θα πρέπει να το κοιτάξουμε μέσω της προτυποποίησης. Ε, ο τομέας αυτό βέβαια έχει ορισμένους περιορισμούς, εξαρτάται από το, την ποιότητα των πληροφοριών που διαθέτουμε και βεβαίω υπάρχουν και ορισμένα άλλα ζητήματα όπως τα υποπροϊόντα, τα οποία δεν μπορεί να επιλύσει αυτή η δημιουργία προτύπων. Από την άλλη, το θέμα της ε, έμεσης αλλαγής της χρήσης γης μπορεί να ε, έχει αντίκτυπο σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή με τη χρήση βιοκαυσίμων. Ε, αλλά βεβαίω ε, ε, θα τηρήσουμε και την αρχή τη αναλογικότητα. Ε, Συμπεράμε ότι υπάρχουν τέσσερι επιλογέ. Πρώτον, να μην αναλάβουμε δράση προ το παρόν, να εξακολουθούμε να παρακολουθούμε την κατάσταση σε επίπεδο ερευνητικών εξέλιξεων. Δεύτερον, να αυξήσουμε το όριο αποταμίευσης εκπομπών νερού του θερμοκηπίου για όλα τα βιοκαύσιμα, κάτι το οποίο μπορείτε να βρείτε σε όλες τις οδηγίες. Τρίτον, να εξετάσουμε το ενδεχόμενο επιπλέον ε, κριτηρίων προϋποθέσεων βιωσιμότητας. και να εξετάσουμε περισσότερο τι συμβαίνει ε, σε διάφορε περιπτώσει, όπω για παράδειγμα στη Βραζιλία και την Αργεντινή. Και Τέταρτον, να ε, εισαγάγουμε ένα συντελεστή ένα παράγοντα που λαμβάνει υπόψη το τι συμβαίνει ε, με, τις, με τα αποθέματα ζωοτροφών από βιοκαύσιμα. Βεβαίως απαιτείται περαιτέρω δημιουργία προτύπων και πρέπει να το συζητήσουμε με άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να συντάξουμε μια αξιολόγηση αντικτύπου εξετάζοντας αυτές τις τέσσερις εναλλακτικέ. Αυτά κάνουμε λοιπόν προς το παρόν. Είναι περίπλοκο το σύστημα όπως ανέφερα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε μια στενή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών μας και εξακολουθούμε ε, να εργαζόμαστε για αυτό την αξιολόγηση αντικτύπου. Έχουμε κάνει πολλά, αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα ε, τη διαδικασία αυτή. Πρώτα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση και εάν είναι απαραίτητο να παρουσιάσουμε μια νομική πράξη. Έχουμε ακόμα δύο μήνες ε, βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχουμε θέσει. Ε, δεν αρνούμε ότι θα είναι πολύ δύσκολο να σας παρουσιάσουμε κάτι μέσα σε δύο μήνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τους κυρίους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις παρουσιάσεις, την παρουσίαση των θέσεων και τις επεξηγήσεις. Να ρωτήσω τους συναδέλφους ποιος θέλει να παρέμβει. Ποιος. Ο κύριος Τόμ ζήτησε τον λόγο. Παρακαλώ κύριε Τόμ, έχετε τον λόγο. Äh, Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, λέει ο κύριος Τούρμες, σε σχέση με την ε, αναδιατύπωση της οδηγίας στην ανανέωση και σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις ε, που είχαμε από τις 12 ως 2 ε, το πρωί, όπου τέλος τέλος καταλήξαμε σε μια συμφωνία που είναι εντολή, νομοθετική εντολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει και να υποβάλει μια πρόταση λύσης για να ληφθεί υπόψη αυτό το στοιχείο την συγκυρία εκείνη και χρονική στιγμή που δέχεται ότι η έμεση αλλαγή χρήσης υπάρχει και είναι σημαντικό στοιχείο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται δεκτό. Σε σχέση με τι προφορικέ τοποθετήσει και διευκρινήσει των δύο εκπροσώπων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως αναφέρθηκε υπάρχει η έμεση αλλαγή χρήσης γης. Εντάξει, υφίσταται αυτό το γεγονός. Λέει λοιπόν με άλλα λόγια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι ένας παράγοντας, ένας συντελεστής σοβαρός αυτό το στοιχείο. Και δεύτερο, λέει ο κύριος Όουεν ότι εντάξει είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, όμως ασχολούμαστε με άλλα θέματα τυποποίησης και υποβολής προτάσεων και όχι μόνο με αυτό όλες οι προβλέψεις σε σχέση με τα θέματα ενέργειας βρίσκονται μέσα σε ένα ρευστό πλαίσιο και φυσικά υπάρχουν αβεβαιότητες όταν έχουμε τέτοια θέματα τυποποίηση. Όλοι γνωρίζουμε όμως ότι υπό τη συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει να δούμε με την αρχή της πρόνοιας, πρόληψης, προφύλαξης precautionary principle. Ακόμα και αν γνωρίζουμε ότι μπορούν να βελτιωθούν τα πρότυπα, αυτό δεν είναι λόγος να μην καταλήγουμε σε απόφαση, σε λήψη απόφασης. Λοιπόν, με άλλα λόγια, γιατί υπογραμμίζω αυτά τα δύο θέματα ξεχωριστά. Αυτό γίνεται επειδή εξακολουθώ να έχω την εντύπωση που έχω αποκομίσει ότι βασιζόμενοι στην ίδια την πραγματικότητα και ιδιαίτερα η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας που ήταν πάντα είχε α, α, κάποιες αντιστάσεις να δεχθούν το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου στο τέλος της διαπραγμάτευσης έχουμε τις κυβερνήσεις ε, και το Κοινοβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο, εμπιστευθήκαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμείς ότι θα προχωρούσε πραγματικά και θα προήγε αυτή την ε, υλοποίηση της νομοθετικής εντολής και θα διευθετούσε τα πράγματα. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν δυσκολίες για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει. Όχι ακριβώς. Και από την άλλη πλευρά έχουμε αρκετά τεκμήρια από τις μελέτες που έχουν γίνει ότι είναι, δημιουργεί πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις η αλλαγή χρήσης γης και έχουμε και πρότυπα, αλλά πρέπει να υπάρχουν άλλοι λόγοι, πολιτικοί λόγοι, ίσως λόγοι που έχει δυσκολίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποδεχθεί το τι γίνεται δηλαδή σε σχέση με κάποια χρόνια πριν και το τι συμβαίνει σήμερα. Όλα αυτά είναι λόγοι για μένα προσωπικά σαν άνθρωπο που διαπραγματεύτηκε όλα αυτά τα θέματα, δημιουργούν δυσχέρειες. Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να δώσουμε εντολή όταν δημιουργείται η εντύπωση στη συνέχεια υστερότερα ότι για κάποιους μη κατανοητού σκοτεινού λόγου δεν μπορεί να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν κάνει τίποτα. Γνωρίζουμε επίση από φήμε ψιθύρους που κυκλοφορούν στου διαδρόμου ότι πιέζει πράγματι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αύξηση των κατοφλίων Όλα αυτά θα σήμαιναν ότι έχει κάποιος αυτοκίνητο χωρίς φρένα και θα έλεγε δεν θα επιδιορθώσω τα φρένα στο αυτοκίνητό μου αλλά θα βελτιώσω το σκελετό του αυτοκινήτου μου ώστε αν χτυπήσει, που θα χτυπήσει και το ξέρουμε και συγκρουστεί με κάποιο άλλο ή με κάποιο τείχο να αντέξει χωρίς φρένα όμως λοιπόν εξακολουθώ να είμαι απόλυτα πεισμένος ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε σχέση με την προτυποποίηση, τα πρότυπα και τυποποίηση. Είναι αυτά τα οποία εμείς ψηφίσαμε στην έκθεση του Κοινοβουλίου, ψηφίσαμε το 2008 και αυτό πρέπει να προαχθεί. Μία λοιπόν εξειδικευμένη επακριβώς ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι η εξής. Για ποιο λόγο, τι συμβαίνει ποιοι είναι οι πολιτικοί λόγοι, τα αίτια για τα οποία έχετε τέτοιες δυσκολίες να προχωρήσετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προαγάγετε αυτά που εμείς θεωρούμε ότι θα έπρεπε να προαχθούν και να υλοποιηθούν με το συγκεκριμένο τρόπο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα το συντελεστή I-Factor με βάση τύπους ε, πρότυπα από πλευράς της Επιστημονικής ε, Επιτροπής Καλιφορνίας που αναθεωρείται και μια και πρέπει να υπάρξουν διορθώσεις, προσωπικά δεν κατανοώ γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τόσες δυσκολίες να το δεχτεί και να υποβάλει μια πρόταση ώστε να ρυθμιστεί αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Έχουμε τέσσερις που έχουν ζητήσει ακόμα τον λόγο. Παρακαλώ τους συναδέλφους να είναι συντομότεροι, γιατί δεν τα καταφέρουμε αλλιώς. Έχουμε και άλλο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ο Πέτρα Λίζα επόμενος, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ. Φυσικά, το Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορεί να το δεχτεί όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συγκεκριμένη εντολή και δεν την υλοποιεί. Απαράδεκτο αυτό και μάλιστα στο νομοθετικό μας έργο από κοινού με το Συμβούλιο, αυτά πρέπει να προχωρήσουν. Παρακαλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γοργά και αποτελεσματικά να εργαστεί. Δεν είμαι όμως απόλυτα πεισμένος ότι είναι η εναλλακτική λύση τέσσερα εκείνη που θα έπρεπε να ακολουθήσουμε. Μια έντονη ίσως και διαφοροποιημένη και γραφειοκρατική θα έλεγα κιόλα προσέγγιση. Εγώ θα ήθελα τρεις ερωτήσεις και πάλι να διατυπώσω που θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Είναι σαφές ότι υπάρχουν ακραίες επιπτώσεις όταν έχουμε αποψήλωση τροπικών δασών, όταν έχουμε ελαιούχους σπόρους, ε, ελε, ελαιοπαραγωγά, φυτά τα οποία καλλιεργούνται εκεί για, βιοκαλλιε... για βιοκαύσιμα και όταν έχουμε την αποψήλωση αυτών των ε, δασών και διαπιστώνεται. Όλα αυτά πρέπει κάπου να συνυπολογίζονται. Υπό το δικό μου πρίσμα δεν μπορούμε να πάμε στο πέμπτο ε, ή δέκατο δεκαδικό στοιχείο μετά την ε, διαστολή, διότι διαφορετικά την υποδιαστολή, διότι έχουμε σε σχέση με τα βιοκαύσιμα και θετικές επιπτώσεις στο κλίμα και πρέπει να προσέξουμε να προχωρήσουμε όμως ε, όταν υπάρχουν, δεν είναι καλής ποιότητας τότε πρέπει να αποφεύγονται και σε σχέση με το συνδυασμό με άλλες επιπτώσεις και σε άλλα θέματα σχετικά πρέπει να ε, υπάρχουν εξετάσεις και έρευνες. Όλοι συμφωνούν ότι υπό το πρίσμα της προστασίας του περιβάλλοντος και για τις πρώτες ύλες πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη καλλιέργεια δασών. Ε, όταν αρχίζουμε τώρα να συζητάμε για τις ε, καλλιέργειες αυτές εκεί όπου ξυλία προηγούμενα υπήρχε πρέπει να δούμε ποιες είναι οι έμεσες επιπτώσεις εκεί όπου για παράδειγμα υπάρχει, υπήρχε δάσος να καλλιεργούνται τρόφιμα ή βιοκαλλιέργειες. Όλοι είμαστε υπέρ για τέτοιες πρωτοβουλίες, αλλά ανά εκτάριο καλλιεργούνται περισσότερα τρόφιμα αν ακολουθεί κανείς ε, τις συμβατικές ε, γεωργικές μεθόδους. Και εδώ υπάρχει συνδυασμός μεταξύ περιβαλλοντικών, ε, επισητιστικών και ενεργειακών παραγόντων. Και είχε γίνει ο και μου είπαν ότι με την ε, αλλαγή την ενεργειακή στη Γερμανία θα χρειαζόμαστε περισσότερες εκτάσεις και αυτό θα έχει μεγάλες επιπτώσεις στην ε, γεωργία. Δεν το είχα σκεφτεί ε, για την αιωλική ενέργεια και το ποσοστό της ε, κάτι τέτοιο σε σχέση με τη γεωργία μας. Έμεσες επιπτώσεις έχουμε παντού και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στα αυτά, σε αυτά που κάνουμε. Πρέπει να υποβάλει κάποια πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να ασχοληθεί με τα ουσιοδέστερα και όχι με τα ε, με μικρολεπτομέρειες και για τα βιοκαύσιμα να μην καταλήξουμε στις αρνητικές επιπτώσεις και έτσι στο τέλος τέλος θα είχαμε θετικές επιπτώσεις αν προσέχαμε το τι θα κάνουμε. Δεν πρέπει υπερβολικά να επιβαρύνουμε γραφειοκρατικά αυτές τις διεργασίες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ Πέτρα Λίζα. Η κυρία Μακάβαν έχει τον λόγο, παρακαλώ. Θα είμαι σύντομη, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα ήθελα να πω ότι δεν ζηλεύω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο η νομοθετική πρόβλεψη προσπαθεί να διακρίνει ανάμεσα στα καλά και στα κακά βιοκαύσιμα. Αυτό ήδη είναι προβληματικό και προσπαθούμε να βρούμε μια λύση. Είναι προφανές ότι υπάρχουν κακά βιοκαύσιμα. Ακούσαμε μια περίπτωση στην Ανατολική Αφρική όπου θα καταστραφεί ένα δάσος για να υπάρξει παραγωγή βιοκαυσίμων για μια Ιταλική εταιρεία, ο κόσμος θα εκτοπιστεί ουσιαστικά από εκεί σε ένα από τους πιο φτωχούς τόπους του πλανήτη. Αυτό πραγματικά γελιοποιεί την περιβαλλοντική μας νομοθεσία, την αναπτυξιακή μας νομοθεσία και αν επιτρέψουμε τέτοιου είδους προγράμματα να ακαποφορήσουν αυτό είναι απαράδεκτο. Αυτό δεν είναι βέβαια μια, παρά μόνο μια άμεση μορφή χρήσης γης. Αλλά το θέμα είναι να προσπαθήσουμε να δούμε αν μια εταιρεία, ένας επιχειρηματίας αγοράσει εδάφη γεωργικά σε μια χώρα στην Αφρική και στο τέλος βλέπουμε ότι καταστρέφεται το δάσος. Αυτό είναι απαράδεκτο. Οι λαοί δεν είναι ισότιμοι σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Κάποιες κοινότητες είναι δύσκολο να διαπραγματευτούν με μεγάλες επιχειρήσεις. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια λύση. Ταυτόχρονα δεν θα ήθελα να σταματήσουμε το σύνολο των βιοκαυσίμων. Δεν συμφωνώ για αυτήν την αντίληψη. Έχουμε ήδη πάντως καθυστερήσει. Ήδη βλέπουμε η έρευνα, οι επενδύσεις στην έρευνα να χάνονται και γι' αυτό θα πρέπει γρήγορα να προχωρήσει η Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σασένης, παρακαλώ επόμενος. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως ο κύριος Τούρμες, ο κύριος Λίζε προανέφεραν, το πόσο αξιό, αξιόπιστη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή και πρέπει να δούμε ότι αυτό δεν αφορά τόσο την Γενική Διεύθυνση για το Κλίμα, αλλά την Γενική Διεύθυνση για τα θέματα ενέργειας που έχει κάποιες αντιστάσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν μελέτες και πρέπει να προχωρήσουμε. Έχει ε, τρεις μελέτες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έδωσε προς σύνταξη και από μία τουλάχιστον του, του Διεθνούς Ινστιτούτου ε, για τις ε, πολιτικές αυτές έρευνες γνωρίζουμε ότι η, τα ηλιοτρόπια, η, η, σόγια και οι άλλες καλλιέργειες ε, δεν ε, ε, συνάδουν με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές για τις, τα ανανεώσιμα. Δεν έχουμε 50% λοιπόν εξοικονόμηση όσον αφορά την χρήση ορυκτών καυσίμων. Αν λοιπόν δεν ληφθούν όλα αυτά, δεν συνυπολογιστούν όλα αυτά και δεν ληφθούν υπόψη σε σχέση με τα βιοκαύσιμα, διακυβεύεται σε σχέση με τις εκτιμήσεις αυτών των μελετών και με βάση αυτές θα είναι σαν να μην λάβουμε υπόψη 14 έως 29 εκατομμύρια επιπρόσθετα οχήματα στην Ευρώπη για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Αυτό είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό και βαρύνο στοιχείο και φυσικά υπάρχει εναλλακτική δυνατότητα και θα πρέπει να ε, ληφθεί υπόψη. Ο κύριος Τουρμέσα ε, τοποθετήθηκε επ' αυτού και πρέπει να περάσουμε στην εναλλακτική δυνατότητα 4. Δηλαδή, ε, σε σχέση με τους συντελεστές ILOC factors, ώστε να μπορέσουμε να διαφοροποιήσουμε τις διαφορετικές εναλλακτικές δυνατότητες σε σχέση με τα βιοκαύσιμα είναι καλά τα βιοκαύσιμα, αλλά να λάβουμε υπόψη και τις διακοιμάσεις αυτές που προανέφερα, να μην τις αγνοήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ούτσακ είναι ο επόμενος αγορητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ένα ερώτημα θα ήθελα να θέσω. Και eh, ε, Νομικού χαρακτήρα. Αναφέρεται στην εμπειρία την οποία είχαμε εδώ και δύο εβδομάδες όταν στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου εγκρίναμε την πρόταση του κυρίου Κρήτον Αρσένη για τα δάση. Με αφορμή αυτή τη συζήτηση είχε τεθεί ένα ερώτημα σχετικό με την εφαρμογή των συνθήκων και της αρχής της επικουρικότητας ακούστηκε ότι ο προορισμός της χρήσης των γεών είναι, των εδαφών είναι εθνική αρμοδιότητα. Εάν εμείς σήμερα λοιπόν εφαρμόσουμε ή προχωρήσουμε προς μια κοινοτική δράση η οποία επιβάλλει δεσμεύσει στα κράτη-μέλη, ποια θα είναι η βασική αρχή την οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να δεσμεύσουμε τα κράτη-μέλη να ακολουθήσουν μια βασική αρχή μια συνεκτική αρχή με αυτά τα οποία είπε η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της σύμφωνη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τρεμόπουλος, τελευταίος αγορητής. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, προφανώς το θέμα έπρεπε να το δούμε σε βάθος, ε, γιατί ακούσαμε για τις επιπτώσεις ε, στα δάση. Υπάρχουν και έμεσες επιπτώσεις. Ε, καλλιεργήσιμη γη που χρησιμοποιείται για παραγωγή τροφίμων μετατρέπεται σε γη για παραγωγή βιοκαυσίμων με αποτέλεσμα να μεταφέρεται έμεσα η καλλιέργεια σε άλλες περιοχές που ήταν ε, βιότοποι. Απελευθερώνονται δηλαδή έτσι τεράστιες ποσότητες διοξίδιου του άνθρακα που ήταν αποθηκευμένες στο βιότοπο, χάνεται φυσικά η βιοπικιλότητα, αποψηλώνεται το δάσος. Τα σχέδια ε, που υπάρχουν για την αύξηση της χρήσης των βιοκαυσίμων στην Ευρώπη την επόμενη δεκαετία απαιτούν παγκοσμίω 69.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα νέων εκτάσεων για τέτοιες ενεργειακές ε, καλλιέργειες και επιδεινώνουν ε, την κλιματική αλλαγή. Υπάρχει αυτή η έρευνα του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής ε, Πολιτικής που μας δίνει πολύ σημαντικά στοιχεία από τη χρήση των βιοκαυσίμων μέχρι το 2020. Ε, λέει λοιπόν ότι ε, η έρευνα αυτή ότι μια περιοχή με έκταση διπλάσια του Βελγίου θα μετατραπεί σε φυτίες και καλλιέργειες λόγω της αναμενόμενης αύξησης ε, στην κατανάλωση βιοκαυσίμων. Αυτή η εξέλιξη θα αυξήσει τις αιτήσει εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 27 με 56 εκατομμύρια τόνους. Αυτό είναι που ε, είπε και πριν ο Κρήτον ότι ισοδυναμεί με την προσθήκη επιπλέον 12 με 26 εκατομμύρια αυτοκινήτων στους δρόμους Ευρώπης ως το 2020. Απαράδεκτο. Στηρίζουμε λοιπόν τα αιτήματα των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Η Επιτροπή θα πρέπει να ανταποκριθεί στο χρονοδιάγραμμα και να εκδώσει μια πρόταση για αυτές τις έμεσες αλλαγές των χρήσεων γης με συγκεκριμένους παράγοντες για τα διαφορετικά είδη βιοκαυσίμων, δηλαδή το option 4. Κύριε Σέμπερ, αυτό είναι ο τελευταίο ίστατο ομιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σωστά δρά όταν με τέτοια προσοχή προχωρεί και θέλω να αναγνωρίσω αυτό το γεγονός και να πω το εκτιμώ, διότι όταν συζητούμε τέτοια θέματα όπως παράγοντες ILOC, βρισκόμαστε σε ένα ανασφαλές επιστημονικά πεδίο, παρθένο πεδίο και όταν έχει δοθεί η εντολή να ληφθεί υπόψη και να εξεταστεί αυτός ο παράγοντας σε σχέση με τις προτάσεις, καλό είναι να είναι κανείς προς προσεκτικός και σε πιστικά αποδεδειγμένα τεκμήρια να βασίζεται. Εδώ κινούμαστε σε ένα τομέα όπου όχι μόνο οι άμεσες αλλά και οι έμεσες επιπτώσεις προέρχονται από αυτόν και θέλουμε να δούμε στην νομοθεσία που θα ε, προταθεί νομοθετικά να ληφθούν όλα αυτά υπόψη γιατί εύκολα μπορεί να δημιουργηθεί παρεμπόδιση και να δημιουργηθούν εμπόδια αν δεν είμαστε συνετοί. Πρέπει να δοθεί ο χρόνος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι συνετή και πρέπει ως Ευρωκοινοβούλιο να μην υπερβιαστούμε και ξεπεράσουμε τη σωστή ε, διεργασία και σωστό ρυθμό, διότι έχει νόημα να ακολουθήσουμε αυτή την αντιμετώπιση σε σχέση με τα ε, βιοκαύσιμα. Αλλά οι έμεσες ε, επιπτώσεις και η ποσοστοποίηση, η εκτίμησή τους με σωστό τρόπο πρέπει να έχει και ένα σωστό επαρκές χρονικό διάστημα για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων, επειδή δεν είναι εύκολη η διαπίστωση όπως στα, στα άμεσα στοιχεία, στις άμεσες επιπτώσεις. Στις έμεσες είναι πιο περίπλοκα τα πράγματα. Πρέπει λοιπόν να μπορέσει να έχει η Επιτροπή το χρόνο να κάνει τη δουλειά. έχω μια μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης για Εσωτερικές Πολιτικές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα έπρεπε ίσως και αυτή να συζητηθεί και να εξεταστεί. Διότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να ληφθεί υπόψη ε, ίσως να προσκληθούν οι συντάκτες αυτής της μελέτης να επεξηγήσουν κάποια πράγματα. Ποιες ε, ποιοι συγκεκριμένοι λόγοι ε, ισχύουν για ε, την στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή τις, ε, τα όσα γύρουν εκείνη ως επιχειρήματα. Ευχαριστώ. Θα δώσω τον λόγο σύντομα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να ολοκληρώσει με την τοποθέτησή της γιατί έχουμε ένα σημείο ακόμα στην ημέρησια αδιάταξη. Θέλω όμως να πω το εξή. Έχουμε και τη Γενική Διεύθυνση για το κλίμα, για τις, τα κλιματικά θέματα. Έχουμε και την Γενική Διεύθυνση σε σχέση με τα θέματα ενέργειας που πρέπει να ληφθεί υπόψη Παρακαλώ, μπορείτε να παρέμβετε. Um, Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω εγώ και σίγουρα ο Χάνς ε, θα συμπληρώσει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι όλοι έχουμε ανάγκη τα βιοκαύσιμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Το ανέφερε σύμφωνα και η Επιτροπή στον οδικό χάρτη για το 2050. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε τα βιοκαύσιμα. Κανείς δεν λέει το αντίθετο θα εξακολουθήσουμε να τα χρειαζόμαστε και στο μέλλον. Επίσης, γνωρίζουμε ότι η δημιουργία προτύπων ε, ε, χρησιμοποιείται ε, ευρέως στην Επιτροπή για την ανάπτυξη πολιτικών, πάντα όμως μα παρουσιάζουν περιορισμούς και συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε την δημιουργία προτύπων όχι για την δημιουργία πολιτικής, αλλά για την ομοθεσία. Έτσι πάμε ένα βήμα παραπέρα και πρέπει να είμαστε σίγουροι τι ακριβώς κάνουμε. Επιπλέον θα σημειώνω αυτά που είπαν ορισμένοι ομιλητέ, που είπαν δηλαδή ότι πρέπει να το κάνουμε σωστά. Αυτό αναφέρθηκε και τον προηγούμενο Νοέμβριο. Καλύτερα είναι να καθυστερήσουμε λίγο, αλλά να έχουμε μια αξιόπιστη και σωστή απάντηση. Αυτό βεβαίω προσπαθούμε και εμεί να κάνουμε. Ε, συζητούμε αυτές τις εναλλακτικές λύσεις ε, στο εσωτερικό της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Γενική ε, γεωργίας, εμπορίου, επιχειρήσεων, όλες αυτές συμμετέχουν. Εξετάζουμε λοιπόν τις αναλυτικές λύσεις όσο δυνατόν πιο επισταμένα. Ωστόσο, όταν ολοκληρώσουμε ε, την εκτίμηση αντικτύπου, η τελική απόφαση θα ληφθεί βάσει πολιτικής συζήτησης. Θα δείσω τώρα το λόγο στον συνάδελφο Χάνς. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Ξέρω ότι θέλετε να κλείσουμε αυτό το σημείο. Έγιναν ορισμένε παρατηρήσει που υπονοούν ότι η Γενική Διεύθυνση Ενέργεια είναι αντίθετη στου ε, συντελεστέ ILOC. Εγώ μπορώ να σα πω ότι αυτό δεν ισχύει. Κανεί δεν έχει λάβει κάποια απόφαση πριν την εξαγωγή αξιολόγηση αντικτύπου. Γι' αυτό ακριβώ την κάνουμε την αξιολόγηση αντικτύπου. Θέλουμε να γνωρίζουμε τον ακριβή αντίκταπο ε, τη μία ή τη άλλη εναλλακτική. Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα σε συμπεράσματα. Ανε, ανεξάρτητα από τις φήμες που μπορεί να κυκλοφορούν από αυτού. Κάτι που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι ο κύριος στόχος της οδηγίας και της ε, ΑΕΠ, ΑΠΕ, συγγνώμη, είναι να δημιουργηθεί αυτή η σταθερότητα και η προβλεψιμότητα, ένα σωστό κλίμα για τις επενδύσεις για όσους θα επενδύσουν σε αυτόν τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Συμφωνούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί ε, γρήγορα αυτό το σημείο, θα πρέπει να βρούμε μια λύση που θα ε, επιλύσει αυτά τα, προβλήματά μας και έτσι οι επενδυτές που επενδύουν σε άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα γνωρίζουν το ρυθμιστικό πλαίσιο. Επιβεβαιώνω λοιπόν τα όσα λέει ο Φίλιπ. Εργαζόμαστε σκληρά, όχι νυχθημερών, αλλά ε, όσο μπορούμε περισσότερο για να ε, κλείσουμε αυτό το φάκελο, ενδεχομένως και ελπίζουμε πριν από το... τις καλοκαιρινές δικοπές. Σας, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και για τη συζήτηση. Και θα δοθεί συνέχεια, δεν υπάρχει τίποτα καθοριστικό. Σας ευχαριστούμε για αυτό. Περνάμε στο τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη, το σημείο 21. Παρουσίαση της μελέτης για τις εκπομπές ε, ρήπων διοξιδίου του άνθρακα από την ΕΜΑΣ. Έχετε τον λόγο για την επόμενη μισή ώρα για να χρησιμοποιήσουμε με το βέλτιστο τρόπο τον χρόνο μας. Παρακαλώ. Αγαπητά μέλη, είμαι συντονιστής εμάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση στη συνάντησή σας και να σας παρουσιάσω τη μελέτη μας για το σύστημα των αντισταθμισμάτων που συνετάχθη από τον παρακαθήμενό μου. Να σας εξηγήσω λίγο ότι το 2008 παρουσιάσαμε μία μελέτη για το ίχνος του άνθρακα, ήταν το πρώτο βήμα για να μειώσουμε τις ε, εκπομπές μας. Σήμερα είμαστε εδώ για να σας παρουσιάσουμε μια άλλη μελέτη η οποία αφορά το σύστημα αντισταθμίσεων διοξιδίου του άνθρακα. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς σαν κοινοβούλιο ε, να προχωρήσουμε σε αυτή την αντιστάθμιση και ποιες είναι οι επιλογές. Το Προεδρείο αποφάσισε να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα μείωσης. Ο σύμβουλος που έχουμε μαζί μας θα σας εξηγήσει τον ρόλο που μπορεί να παίξει το offsetting σε αυτή την προσπάθεια. η μελέτη έγινε από την εταιρεία Deloitte, από τον κύριο Τιμπό και από έναν άλλο σύμβουλο. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Μετά από την παρουσίαση θα είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Hello. Ευχαριστούμε που μας δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα σχετικά με τις αντισταθμίσεις των εκπομπών που εκπέμπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να ενθυμίστε ότι στόχος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η μείωση του ίχνου σε άνθρακα 20% από το 2006 μέχρι το 2020. Το 2008 κάναμε μια μελέτη για το ίχνος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ίχνος σε άνθρακα και προτείναμε τη μείωση κατά 30%. Το πρόγραμμα δράσης έγινε δεκτό από το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Φεβρουάριο του 2009 και συμπεριελήφθη στο πρόγραμμα δράσης ΕΜΑΣ. Στόχος του προγράμματος εμάς ήταν να γίνει μια μελέτη των εκπομπών τις οποίες παράγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι περιλαμβάνει λοιπόν το ίχνος άνθρακα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στη λήψη πολλών μέτρων. Καταρχάς, έχουμε τις εκπομπές ε, οι οποίες παράγονται από ρηκτά καύσιμα για τη θέρμανση και τον κλιματισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης τα συστήματα ψήξης, την ενέργεια που χρησιμοποιείται για τις μεταφορές, τις μεταφορές ε, υπαλλήλων, μελών, επισκεπτών, οι πτήσεις από τις ε, ε, διάφορες χώρες προς τις Βρυξέλλες και το Στρασβούργο δεν περιλαμβάνονται στο υπολογιστέν μέχρι τώρα ίχνος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και προσπαθήσαμε επίσης να δούμε και το ίχνος το οποίο προκαλείται από τους προμηθευτές, από τον εξοπλισμό Η μελέτη που κάναμε άλλωστε έχει και αυτή καταναλώσει ε, διοξίδιο του ανθρακά. Αν και το πρόγραμμα το οποίο προτείνουμε είναι ουδέτερο σε επίπεδο εκπομπών. Επίσης αναφερόμαστε και στην, στο ίχνος το οποίο παράγεται από τις κατασκευές, τις οικοδομικές δραστηριότητες, τις επισκευές κτλ το οποίο προσπαθούμε να εξισώσουμε, να ισορροπήσουμε και να αποσβέσουμε κατά τη διάρκεια της περίοδου λειτουργίας του προγράμματος. Προσπαθούμε να βελτιώσουμε επίσης την κατάσταση και σε όλους τους τομείς στους οποίους μπορούμε να επηρεάσουμε εξωτερικά, όπως κατασκευαστές, παροχής υπηρεσιών στον τομέα της εστίασης κτλ. Βασισμένοι λοιπόν στα στοιχεία που συλλέξαμε από το 2006 έχουμε κάποια πρώτα θετικά στοιχεία. Τα πράγματα εξελίχθηκαν θετικά από τότε. Έχουμε μία μείωση 14% ανά υπάλληλο. Οι πιο σημαντικές εκπομπές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλονται στις μεταφορές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν είναι στην πορεία να πετύχει τους στόχους του 30% και το θέμα είναι τι μπορούμε να κάνουμε με το υπόλοιπο 17%. Εδώ το offsetting, οι αντισταθμίσεις μπορεί να παίξουν κάποιο σημαντικό ρόλο. Η μελέτη λοιπόν έχει σαν στόχο την ανάλυση του τι θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον περίμετρο offset του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι εννοούμε γι' αυτό. βασικός στόχος είναι να διαφοροποιήσουμε τα διάφορα συστήματα τα οποία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ή για να προχωρήσουμε στην αντιστάθμιση. Πώς θα το κάνουμε αυτό, να αναλύσουμε τις μεθόδους που θα ακολουθήσουμε και να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια και την αξιοπιστία των διαδικασιών αντιστάθμισης. Η διαδικασία αυτή ε, ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια. Τα πρώτα τρία στάδια έγιναν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη. Μετρήσαμε λοιπόν τα ίχνη άνθρακα, τις εφαρμοστές στρατηγικές και τώρα ε, επαναυπολογίσαμε τα αποτελέσματα των εφαρμοσμένων στρατηγικών και ήδη έχουμε όπως είπαμε μία κάποια μείωση. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε λοιπόν με το υπόλοιπο 70%. Και εδώ όπως είπαμε η αντιστάθμιση μπορεί να παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο. Οι μειώσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να στηρίξουμε ε, προγράμματα όπως στην Αφρική Έτσι θα μπορούσαμε λοιπόν εν μέρη το κομμάτι του 70% να το αντισταθμίσουμε με αφρικανικές χώρες και έτσι το Κοινοβούλιο θα αναλάβει τις ευθύνες του για τις υπόλοιπες αυτές εκπομπές. Um, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα επαληθεύσιμα προγράμματα που μειώνουν τις ε, εκπομπές. Τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να πιστοποιηθούν από αναγνωρισμένες αρχές έτσι ώστε η αξιοπιστία τους να είναι δεδομένη και τα προγράμματα να είναι πράγματι υπαρκτά. Αυτό θα μεταφερθούν τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας στους λογαριασμούς ITL, τους οποίους έχει το Κοινοβούλιο. Και η οικονομική στήριξη θα πρέπει να συνεχιστεί θέτοντας χρηματοδότες όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε επαφή με αυτούς που θα είναι υπεύθυνοι για τα προγράμματα στην Αφρική. Αυτό σημαίνει ότι θα πάρουμε πιστοποιητικά για τις, ε, για τις εκπομπές οι οποίες γίνονται σε άλλη χώρα που είναι ισότιμα σε επίπεδο εκπομπών με τις μειώσεις τις οποίες κάνουμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι αντισταθμίσεις αυτές δεν θα χρησιμοποιούνται, δεν θα χρησιμοποιούνται συγγνώμη, από τρίτα μέρη. Αυτά είναι όχι προτάσεις αλλά παραδείγματα για το τι είδους προγράμματα αυτή η χρηματοδότηση της αντιστάθμισης θα μπορούσε να στηρίξει. Υπάρχουν προγράμματα βιομάζας, παραγωγής βιομάζας στην Αφρική. Η βιομάζα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αντικατάστασης ε, ε, ορυκτών καυσίμων όπως γεννητριών με ε, πετρέλαιο αιωλικά επίσης συστήματα παραγωγής, ένταξη στο δίκτυο της παραγωγής από αιωλική ενέργεια και αντικατάσταση παραγόμενων ποσοτήτων ηλεκτρισμού από ορυκτά καύσιμα όπως άνθρακα. Επίσης και αντικατάσταση του μεθανίου που παράγεται από τις χωματερές σε χώρες όπως η Τανζανία και έτσι μπορούμε να μειώσουμε τους κινδύνους που υπάρχουν, τις ασθένειες που προκαλούνται και την άσχημη μυρωδιά. Αυτή η προσπάθεια όμως παράγει βέβαια αέρια του θερμοκηπίου. Υπάρχουν επίσης και ηλιακά πάνελ, ηλιακοί πίνακες στην Νότιο Αφρική που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την θέρμανση και τον κλιματισμό οικειών στην περιοχή. Το θέμα είναι ότι αν ακολουθήσουμε αυτήν την πορεία, τι μπορούμε να αντισταθμίσουμε. Και εδώ γίνεται η πρόταση. Οι πτήσει, όπως είπαμε, που οδηγούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τώρα. Γι' αυτό θα πρέπει να προσωπολογιστούν και κάθε Ευρωβουλευτής θα μπορεί να αντισταθμίζει τις πτήσει του ή τις πτήσει της σε εθελοντική βάση. Υπάρχουν τρεις περίμετροι αντισταθμίσεις που ε, ε, περιγράφονται. Πρώτον θα μπορούσαμε μόνο να αντισταθμίσουμε τις πτήσεις του προσωπικού, γιατί πριν μίλησα μόνο για τις πτήσεις των βουλευτών και αυτό θα κοστίσει 108.000 ευρώ κατ' έτος. Το δεύτερο στάδιο, η δεύτερη περίμετρος, θα είναι να αντισταθμίσουμε το σύνολο των ταξιδιών του προσωπικού και την ενέργεια που καταναλώνεται στα κτίρια, ηλεκτρισμό και φυσικό αέριο. Αυτός ο ενδιάμεσος χώρος θα αντικατοπτρίζει 605.000 ευρώ κατ' Η τρίτη μεγαλύτερη περίμετρος θα είναι η αντιστάθμιση του συνόλου του ίχνους που παράγεται από το Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι θα αντισταθμίσουμε όλες τις εκπομπές εκτός των πτήσεων των βουλευτών, όλες τις πτήσεις του προσωπικού, τα κτίρια, τις μεταφορές, τα αυτοκίνητα και υπηρεσίες ε, όπως ε, τα απόβλητα, ε, τα απορρίμματα, ο καθαρισμός, η εστίαση κτλ. Για την αντιστάθμιση όλων αυτών μιλάμε για 2 εκατομμύρια ευρώ κατ' έτος. 20 ευρώ ανατόνο διοξιδίου του άνθρακα. Αυτή είναι λοιπόν η πρόταση την οποία στο Προεδρείο, θα στείλουμε στο Προεδρείο κατά τη διάρκεια του θέρους. Υπάρχουν θέματα με την αξιοπιστία και τα επίπεδα της αντιστάθμισης και εδώ έχουν υπάρξει κάποια προβλήματα και με τα μέσα ενημέρωσης. Το θέμα είναι ότι δεν θα πρέπει τα μέτρα αυτά να βλάπτουν άλλους τομείς και θα πρέπει επίσης να παρέχονται ε, και θετικά, θετικές επιπτώσεις σε κοινωνικο-οικονομικούς τομείς. Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι μερικές φορές ορισμένοι θεωρούν το offsetting, της αντισταθμίσης σαν κάτι το οποίο γίνεται εφάπαξ από εκεί και πέρα έχει κανείς καθαρίσει, έχει ξεμπλέξει. Δεν είναι έτσι. Κάποιοι αναλαμβάνουν τη μείωση των εκπομπών τους και δυστυχώς μετά περνούν σε πλαστές μειώσεις οι οποίες ζητούν να ληφθούν υπόψη πριν από την αντιστάθμιση. Γι' αυτό πρέπει να γίνουν οι μελέτες εκ των προτέρων. Το ίδιο ισχύει και για το ανακυκλωμένο χαρτί το οποίο χρησιμοποιείται. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, ότι αυτός ε, που χρησιμοποιεί το ανακυκλωμένο χαρτί μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερο γιατί προέρχεται από μια σωστότερη πηγή. Αυτό το οποίο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή μειώσει το χαρτί σου, χρησιμοποιείς και ανακυκλωμένο χαρτί επιπλέον. Και εδώ λοιπόν θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε την παραγωγή εκπομπών και τότε θα περάσουμε στην αντιστάθμιση. Στη διαφάνεια βλέπετε κάποια παραδείγματα για τα επίπεδα τα οποία υπάρχουν. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ληφθούν υπόψη. Εμείς συστήνουμε στη μελέτη αυτή οι μηχανισμοί καθαρής ανάπτυξης να χρησιμοποιούνται όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα ETS Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει δεκτό από τις οργανώσεις αυτές και είναι λογικό να χρησιμοποιηθεί ε, εκ νέου και στα πλαίσια της εθελοντικής αντιστάθμισης από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ανιχνευσιμότητα των αντισταθμίσεων αυτών είναι σημαντική για να δείξουμε ακριβώς τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η φάση στην οποία υποστηρίζεται το πρόγραμμα είναι επίσης σημαντική. Πρέπει να υποστηρίξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο δημιουργεί διαδραστικές αντιδράσεις, οι οποίες όμως θα πρέπει να αποφευκτούν μερικές φορές και δεν θα πρέπει εμείς τις μειώσεις αυτές να τις αφαιρέσουμε από προγράμματα τα οποία είναι ήδη σε λειτουργία και να προκαλέσουμε τεχνολογικούς κινδύνους για την εξέλιξη των προγραμμάτων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε ex post τις βεβαιωμένες αντισταθμίσεις. Μία ερώτηση την οποία μπορείτε να θέσετε είναι το τι γίνεται με τις άλλες ε, διοικήσεις γύρω από την υπόθεση αυτή. Έχουμε αναλύσει κάποιες από τις, κάποιους από τους οργανισμούς αυτούς, τα Ηνωμένα Έθνη αντισταθμίζουν την ενέργεια την οποία καταναλώνουν σε επίπεδο ταξιδιού και οικοδομών, ε, προχωρώντας στην ουδετερότητα στον τομέα του άνθρακα. Στη Μεγάλη Βρετανία η Κάτω Βουλή επίσης αντισταθμίζει το σύνολο των αερομεταφορών, το Bundestag επίσης αντισταθμίζει το ίχνος των ταξιδιών, των βουλευτών, των υπουργείων, των υπαλλήλων με ένα προϋπολογισμό 2 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης και άλλα κοινοβούλια, σουηδικά, αμερικανικά, ελβετικά, και αυτοί αντισταθμίζουν το σύνολο των πτήσεών τους και το, την λειτουργία των κτηρίων τους. Επίσης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποιες ε, ε, πολιτικές ομάδες ε, και οι πτήσεις που είχαν κάνει τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Κανκούν έτυχαν αντιστάθμισης. πάρε, Επομένω, τέλο, ε, ποιο θα είναι το όφελο ε, τη συμμετοχή στο Ευρωκοινοβουλίο εδώ πέρα. Δείχνουν έτσι ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για το σύνολο των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Θα αποτελέσει παράδειγμα και πρότυπο για, για τον υπόλοιπο κόσμο και έτσι θα μπορεί να διαδώσει και το ε, μήνυμά του πιο εύκολα. Θα ενισχύσει τη δεσμεύση επίπεδο κλίματο που έχουν γίνει σε διεθνές επίπεδο. Θα πάμε πέρα από το 30% ε, τον στόχο που έχει διαμορφωθεί για την μείωση των εκπομπών. Θέτουμε μια τιμή, ένα κόστος για τον άνθρακα και αυτό λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις ε, ε, αποφάσεις που λαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα λαμβάνω δηλαδή υπόψη τον αντίκτυπο σε επίπεδο διοξιδίου του άνθρακα σε κάθε απόφαση που λαμβάνουν. Ε, στηρίζουμε την ε, οικονομία χαμηλού άνθρακα και στηρίζουμε και άλλες χώρες ε, που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες χωρίς να ξεχνάμε τις δεσμεύσεις που έγιναν στην Κανκούν. Έχει παρουσιαστεί το, το πρότυπο, το παράδειγμα ενός βυθιζόμενου πλοίου όταν πέσει κάπου πάνω το πλοίο, προφανώ και χρειάζεται ε, κάποια μέτρα για να επιλύσει προσωρινά το πρόβλημα. Αυτό είναι το, η μείωση κατά 30% που έχουμε θέσει ω στόχο. Αλλά για το υπόλοιπο 70% ε, μπορούμε να το συγκρίνουμε με το, νερό που, που συνεχίζει και μπαίνει στο πλοίο ενώ εσύ το επισκευάζεις. γιατί επισκευάζεις με τον πλοίο, αλλά πρέπει να πάρεις κουβάδες για να, για να πετάξεις έξω το, το νερό που έχει μπει. Αυτό λοιπόν ε, είναι αναπαριστά το 70% που ε, μας απομένει ακόμα για την επίτευξη των στόχων μας, περιμένοντας όλες αυτές τις τεχνολογίες που θα έρθουν στο μέλλον. Μάλιστα, σα ευχαριστώ λοιπόν θερμότατα για την παρουσίαση, την εισήγηση αυτή. Πρέπει να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν είναι τόσοι πολλοί παρόντες από του ευρωβουλευτέ. Ο συνάδελφο Αρσένη το βρήκε πραγματικά ενδιαφέρον και παρέστη. Κρίμα ότι οι άλλοι δεν παρέστησαν και δεν άκουσαν την ε, εισήγηση. Αλλά θα τα διαβάσουμε αυτά και σίγουρα θα τα διαβάσουν και οι άλλοι. οποίο ε, έχει ε, κάποια ερωτήματα πραγματικά εκπλήσεται όπω και εγώ είναι πραγματικά μεγάλη η εμβέλεια αυτών που μας προτείνεται και εγώ ως ε, υπεύθυνη για τον προϋπολογισμό και τα δημοσιονομικά θα ήθελα να μπορούσαμε να είχαμε τη δική μας εξοικονόμηση εμείς εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο για να μπορέσουμε να εξαγοράσουμε αυτή την ας το πω έτσι υποχρέωσή μας αυτή την, τα βάρη τα οποία ε, έχουμε επομιστεί ε, σε σχέση με μια μεγάλη οργάνωση και τις ε, συστάσεις της. Από ό,τι κατάλαβα, δυστυχώς αυτή είναι η μόνη δυνατότητα. Και αυτό με θλίβει ιδιαίτερα. Θα πίστευα θα μπορούσαμε και τα κλιματιστικά να τα χαμηλώσουμε για να καταφέρουμε κάπως να συνεισφέρουμε. Αλλά αυτό θα ήταν μία, στο πω ε, μία αποτελεσματική παρέμβαση. Εσείς θέλετε να πείτε κάτι. Είμαστε οι μόνοι οι οποίοι είμαστε παρόντες εδώ, δεν υπάρχουν άλλοι. Θέλω να σας δώσω εσά ε, τον λόγο και πάλι. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Κάτι πολύ σημαντικό για μας είναι ότι η αντιστάθμιση αυτή δεν ε, υποκαθιστά την μείωση των εκπομπών διοξυδίου του άνθρακα. Θα εξακολουθήσουμε να μειώνουμε τις εκπομπές μας. Υπάρχει ένα ε, σχέδιο για την μείωση αυτή. Ε, και θέτει αυτό το στόχο το 30%. Ωστόσο, το μόνο που λέμε είναι ότι υπάρχει μια αναλεκτική λύση για το υπόλοιπο 70%. Δεν θα μειώσουμε τι ε, προσπάθειέ μα για την, για μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Θα είναι μια συμπληρωματική προσπάθεια. Ναι, παρακαλώ, εσεί έχετε τον λόγο. Να σα ευχαριστήσω για αυτή την παρουσίαση. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Φυσικά και δεν μπορούμε να ε, υποκαταστήσουμε την μείωση των εκπομπών με το offsetting, την αντιστάθμιση, αλλά το μέσο αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Αν κατάλαβα καλά, το κόστος για το κοινοβούλιο είναι 2,5 δις ευρώ. Καλά το κατάλαβα. Ποιο είναι το εκτιμόμενο κόστος για το κοινοβούλιο. Ναι. Έχουμε ένα σύστημα μεταβλητών που ε, ξεκινά από ένα ελάχιστο ε, σε μέσο ή και ε, ουδέτερος προς τη χρήση άνθρακα. Εκεί πέρα δηλαδή μειώνουμε όλες τις εκπομπές. Και αυτό αυξάνει το κόστος από, τα, από τις 100.000 ευρώ στα 2 εκατομμύρια. Και από αυτά τα 2 εκατομμύρια ποιο είναι το λειτουργικό κόστος των υπηρεσιών και ποιο ποσοστό ε, κατευθείαν ε, στο offsetting, δηλαδή στις αποταμιεύσεις ε, σε, σε του ανθράκα. Τα 2 εκατομμύρια εδώ πέρα σημαίνει ότι υπολογίζουμε το τρέχον ίχνος μας. Μετά έχουμε ε, μια τιμή του, της αγοράς, 20 ευρώ ανατόνο, και έτσι καταλήγουμε στο, στα 2 εκατομμύρια. Δηλαδή κοστολογούμε τις εκπομπές μας. Τις υπολογίζουμε και λέμε με μία μέση τιμή 20 ευρώ τον τόνο φτάνουμε στα 2 εκατομμύρια για να ε, ε, αντισταθμίσουμε όλες τις εκπομπές μας. Δεν έχει σχέση με το λειτουργικό κόστος. Βασίζεται στις εκπομπές μας. Ε, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, είχαμε περίπου 100.000 ε, τόνους διοξιδίου του άνθρακα. Καταλήγουμε επίσης σε μια μέση τιμή 20 ευρώ ανά τόνο και έτσι φτάνουμε στο τελικό ε, αριθμό. Μια τελευταία ερώτηση. Από ό,τι κατάλαβα πρέπει να αγοράσουμε αυτή την ποσότητα διοξιδίου του άνθρακα το, το δικαίωμα που αντιστοιχεί σε αυτό. Αλλά τι θα πρέπει να πληρώσουμε επιπλέον για το λειτουργικό κόστος. Δηλαδή, ποσά που δεν θα διοχετευτούν κατευθείαν για την αποταμίευση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Για την εξοικονόμηση μάλλον εκπομπών να του άνθρακα. Δεν ξέρω αν ήμουν σαφής. Ελπίζω να κατάλαβα το ερώτημά σας. Ε, λέτε, αν μειώσουμε τις εκπομπές, ποιο θα είναι το λειτουργικό κόστος. Ναι, καλύτερα να τα συζητήσουμε μετά, φεύγοντας. Äh λοιπόν, εντάξει, για τις διμερείς ε, συζητήσεις ε, που μπορούν να ακολουθήσουν. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για τα όσα μας είπατε. Πρέπει να παραμείνουμε ακολουθώντας αυτή την πορεία, κάνοντας νέους υπολογισμούς, ε, βλέποντας τι θα κοστίσουν όλα αυτά για την εξοικονόμηση. Αυτό είναι τουλάχιστον αυτό που αποκομίσαμε ως μήνυμα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά. Και ολοκληρώνεται η συζήτηση για απόψε. Θα συνεχίσουμε αύριο στις 9 με τους συντονιστές και στις 10 θα αρχίσει Πάλι η συνεδρίασή μας, η τακτική συνεδρίαση. Καλό βράδυ σε όλους σας. Ευχαριστώ. Γεια σας. <laughs>